συνεχίζουμε με μια μικρή καθυστέρηση για λόγους τεχνικούς και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Υπενθυμίζω να τσεκάρετε αν έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ζητήσετε να σας τη φέρουν την κάρτα αν δεν την έχετε ήδη μαζί σας. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Έχουμε μια πολύ μακρά ημερήσια διάταξη σήμερα. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Και περνώ αμέσως στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας ενημερώνω ότι μετά από έτοιμα της εισηγήτριας κυρίας Χαράνς Γκαρσία, το σημείο 6 για τα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες έχει αναβληθεί για την 5η στις 9 το πρωί. Όπως είπα, αυτό έγινε μετά από αίτημα της εισηγήτριας. Έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίαση τη 7 η Ιουλίου. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θα υποθέσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Ε, η συνεδρίασή μας προβάλλεται στο διαδίκτυο και υπενθυμίζω ότι σήμερα είμαστε εδώ, αύριο όμως θα είμαστε στο Γιάννη 4Q2, έχουμε διερμηνία σε 16 γλώσσες. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης για τον προϋπολογισμό του 2015 που παρουσιάστηκε από τον Πέτερ Γιάρ στις 23 Ιουλίου. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για τη γνωμοδότηση και τα στοιχεία του προϋπολογισμού ήταν 25 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι και λόγω της προεκλογικής περίοδου το χρονοδιάγραμμα ήταν πάρα πολύ στενό και το σχέδιο γνωμοδότησης υπήρχε μόνο στα αγγλικά και οι τροπολογίες μπορούσαν να κατατεθούν μόνο στα αγγλικά. Ελάβαμε 24 ε, τροπολογίες για τη γνωμοδότηση και 66 για τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Κύριε Γιάρ, έχετε το λόγο. Πέτερ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι λόγω των ευρωεκλογών ήταν πολύ στενή η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, όμως τα καταφέραμε. Ευχαριστώ σε αυτό το σημείο όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι λόγω των γεγονότων ε, μας έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις ε, από τότε, από τον Ιούλιο του 2015, αντιμετωπίζουμε στον οπροκυπευτικό τομέα μεγάλη κρίση, καλή συγκομιδή, συνδεδεμένη με το ρωσικό εμπάργο, το οποίο δημιουργεί μεγάλες αναταραχές στον τομέα. Είμαι ευγνώμων στην Κομισιόν που προέβησε άμεση λήψη ε, μέτρων και διάθεσε 125 εκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Όποιοι όμως μπορούν να κάνουν ε, λογαριασμούς, και δουν τα ποσά, τα έχουν μελετήσει και τα έχουν κατανείμει στους τομείς. Όποιος τα ξέρει αυτά βλέπει ότι τα χρήματα δεν θα επαρκέσουν. Παρακαλώ λοιπόν την Επιτροπή μετά την ε, ψηφοφορία στο τέλος να προχωρήσουμε σε κάποιο ψήφισμα ή διατύπωση άποψης λέγοντας ότι γνωρίζουμε ότι και για τη σταθερότητα του προϋπολογισμού ε, εν ώψη αλλαγών. Είμαστε διατεθειμένοι, αν παραστεί ανάγκη, να αυξήσουμε αυτό το Ταμείο για τις Κρίσεις. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει ε, τι θα συμβεί, πάντως θα ψηφίσουμε σήμερα. Και γνωρίζουμε ότι η κρίση υπάρχει, είναι δεδομένη. Αυτό θέλω να δηλώσω. Θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα συγκεκριμένα μετά από μία δήλωση προθέσεων για να στείλουμε και στους συναδέλφους στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι θα υπάρξει συνέχεια εδώ. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, γνώστες της διαδικασίας πώς μπορούμε να μεθοδεύσουμε το θέμα με τον καλύτερο τρόπο, ούτως ώστε να περάσει το μήνυμα αυτής της δήλωσης προθέσεων από την πλευρά μας. Και τώρα κοιτώ το Προεδρείο για να μάθω πώς θα μπορέσουμε να προβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ε, πολιτική δήλωση προθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η δήλωσή σας αλλά και η φύση του προβλήματος ε, είναι κατεπήγοντα θέματα και γι' αυτό ρωτώ ζητώ από τους συναδέλφους στη Γραμματεία να σκεφτούν την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για μια τέτοια δήλωση. Θα ήθελα όμως να επαναλάβετε και επίσημα το έτοιμά σας αυτό μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού για να συμπεριληφθεί στα έγγραφά μας. Και πιστεύω ακόμη ότι το θέμα θα συζητηθεί αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στην ψηφοφορία, εκτός και άποιος ζητεί, αν κάποιος ζητεί το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Κύριος Μπικονού. Ναι, λέγομαι Γουανάνο. Σας ε, υπέβαλα μια τροπολογία για το ρύζι, την οποία θα ήθελα να τροποποιήσω προφορικώς και να είναι λίγο πιο ήπια, για να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για την προάσπιση του ρυζιού, ε, το Ιταλικού προς το παρόν, αλλά προφανώς η τροπολογία αυτή αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβάσω την ε, ε, τροπολογία ώστε να μην υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές ε, για συγκεκριμένες περιοχές. Ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προσέξουν ιδιαίτερα τον τομέα τουρισμού και επισημαίνει τη σημασία της προστασίας των παραγωγών από τις ανισορροπίες αγοράς που ε, προκαλούνται από εισαγωγές ρυζιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσο μπορώ να κάνω αυτή την αλλαγή ε, μέσω αυτής της προφορικής τροπολογίας. E, Νομίζω ότι αυτή η τροπολογία θα ψηφιστεί όταν ε, θα φτάσουμε στην τροπολογία, Επομένω, τότε θα ήθελα να τη διαβάσετε ξανά ω προφορική τροπολογία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο το λόγο, από ό,τι βλέπω όχι. Να ψηφίσουμε λοιπόν Ε, φαντάζομαι ότι έχετε όλοι τις ε, κάρτες σας. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Ερώτηση, παρακαλώ. Δεν έχω την κάρτα. Α, έχω την... έχω την κάρτα μου, αλλά... Α, πάντα την έχω, αυτή τη φορά δεν την έχω. Ε, εντάξει, να δούμε, θα το δούμε μετά, εάν υπάρχουν προβλήματα και αν υπάρχουν διαφορές. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Τροπολογία 53.00 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρασε τη ψηφοφορία. I have Υπάρχει ένας επιπλέον φιλελεύθερος, ένας επιπλέον από το ECR και ένας ε, σοσιαλιστής επιπλέον. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία γιατί έχουμε τρεις επιπλέον ψήφους. Σας παρακαλώ, δείτε λίγο τη σύνθεση των ομάδων σας. Επαναλαμβάνετε ψηφοφορία λοιπόν. Άρχεται ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 5300. Ευχαριστώ. Πέρασε της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έχετε τα αποτελέσματα στην οθόνη σας. Περνάμε λοιπόν τώρα στην 5301. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρασε ψηφοφορία. Και πάλι έχουμε έναν επιπλέον φιλελεύθερο. Επαναλαμβάνεται λοιπόν η 5301. Άρχεται η ψηφοφορία. 5301. Θα ήθελα να ε, λύσουν το θέμα τους όλες οι πολιτικές ομάδες, γιατί έχω και έναν επιπλέον από το ΕΛΚ και έναν επιπλέον ακόμα. Σας παρακαλώ λοιπόν δείτε λίγο τις θητές των ομάδων σας. Σας παρακαλώ λοιπόν επαληθεύστε λίγο τη σύνθεση των ομάδων σας. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Για την 5301 δεν ψηφίζουμε την 5325, αλλά την 5301. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρασε ψηφοφορίας. ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη συνέχεια στην 5302. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρασε της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 5303. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5304. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5305. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέραση ψηφοφορία. Ένας επιπλέον μη εγγεγραμμένος. ούτως ή άλλω δεν είχε μεγάλη σημασία, Επομένω μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, στην επόμενη τροπολογία. Περνάμε λοιπόν στην 5306. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. πέρασε τη ψηφοφορία. Και πάλι έχουμε έναν επιπλέον μη εγγεγραμμένο και πάλι όμως δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. 5361. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5307. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 5308. Ο κύριος Ντες. Ναι κύριε Πρόεδρε, είμαστε 42 μέλη δεν μπορούμε να είμαστε 43. Η μία εγγεγραμμένη μπορεί να είναι μεν μία εγγεγραμμένη, αλλά πρέπει κάπως να συμφωνήσουν γιατί πρέπει να έχουμε σωστό αποτέλεσμα. Είμαστε 42, όχι 43. Ο κύριος ε, Ταραμπέλα λυπάμαι, πρέπει να πω στους μη εγγεγραμμένους, πρέπει να γίνονται σεβαστοί κάποιοι κανόνες, όταν πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες ψήφοι, πρέπει να συγκεκριμένες ψήφοι. Ναι, μεν δεν έχει σημασία για την ε, ψηφοφορία, αλλά σας παρακαλώ να αποσύρετε την επιπλέον, ε, το άτομο το οποίο ψηφίζει επιπλέον, πρέπει να γίνονται σεβαστοί κανόνες. Ναι, πολύ καλά. Όντω οι μη εγγεγραμμένοι μπορεί να μην έχουν μια πολύ συγκεκριμένη δομή, αλλά σας παρακαλώ συνεννοηθείτε για να ξέρετε ποιο ψηφίζει και ποιο όχι. Και να αποφασίσετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν εξ ονόματο ε, αυτών. Κύριε, κύριοι Ντός, Φερό και Γουαζό είναι οι μη εγγεγραμμένοι. Επειδή είναι παρόντες και οι τρεις, είναι κανονικά οι τρεις ε, μη εγγεγραμμένοι που θα πρέπει να ψηφίζουν σήμερα, εκτός ε, και αν θέλετε να πείτε ότι υπάρχει και αναπληρωτές. Τρεις ψήφοι είναι εδώ ε, αποδεκτές, έχουμε και τα τρία τακτικά μέλη παρόντα, επομένως θα πρέπει να ψηφίσετε και εσείς οι τρεις μόνο. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι για αυτή την επίθεση από τον κύριο. Είμαστε τρει ε, μία εγγεγραμμένοι, ψηφίζουμε. Νομίζω ότι πρόκειται για λάθο. Ο κύριο Ταραμπέλα διακόψει. Κοιτάξτε, έχουμε και εμεί ένα πληρωτή εδώ, δεν ψηφίζει, έχουμε και εμεί πειθαρχία στην ομία μα. Είμαστε τρει μία εγγεγραμμένοι από ό,τι γνωρίζω. Ο κύριος Μπονάνο είναι αναπληρωτή και ψηφίζει. Μπορεί να ψηφίζουν και αναπληρωτέ. Πώ ψηφίζει αν δεν έχει κάρτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πώ γίνεται. Με τι κάρτα ψηφίζει. Ε, ε συγγνώμη, ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δούμε τουλάχιστον τι γίνεται, γιατί εγώ διαπιστώνω εδώ ότι υπάρχει μια διάθεση να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι είναι απίθαρχη μια γεγραμμένη και νομίζω ότι θα πρέπει να δείτε πώς ψηφίζουμε αυτής εξ αρχής. Υπάρχει ε, ε κανονισμός ο οποίος προβλέπει ότι πρέπει να ψηφίζουμε ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών. Καταλαβαίνω ότι τώρα που αφηνίστηκαν ε, όλα, αφού ακούσαμε τη γραμματεία και τα μέλη, ελπίζω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα θα είναι σωστή η ψηφοφορία. Ο κύριος Μονάνο, συγγνώμη. Εγώ δεν ξέρω τους κύριους Στατ και Τεραμπέλα. Εγώ ε, Προτάρησε εδώ. Ήρθε εδώ και ρώτησα, μπορώ να ψηφίσω, αν δεν μπορώ να ψηφίσω ζητώ συγγνώμη. Αλλά μια τέτοια συμπεριφορά ενό ατόμου απέναντι σε ένα άλλο άτομο που έρχεται εδώ και είναι ευρωβουλευτή εδώ και λίγε εβδομάδε ε, δεν ε, είναι μια συμπεριφορά αποδεκτή. Καταλάβετε τώρα, εγώ έχω την κάρτα, ε, τι να κάνω να την πετάξω στο πρόσωπο, δεν είναι τώρα αυτή η σωστή συμπεριφορά. Να την πετάξω στο κεφάλι, τι να κάνω. Ναι rozumiemy pana, rozumiemy pana wypowiedź, ale jak znamy pana... Μάλιστα, κατανοούμε τι λέτε. Ξέρουμε βέβαια πολύ καλά τον κύριο Ταραμπέλα, ξέρουμε την προσωπικότητά του. Ζητώ συγγνώμη από εσά και νομίζω τώρα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Και περνάμε στην 5308 αρχή τη ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 5309. Άρχεται ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 5310. Άρχεται ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 53-11. Άρχεται η ψηφοφορία για την 53-11. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53-62. Άρχεται η ψηφοφορία. 53-62. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53-12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. Τροπολογία 53, 13. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 53, 55. Άρχεται η ψηφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία Τροπολογία 53-14. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 53-15. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ εγκρινεται Εγκρίνεται. 5316 53-16. Άρχεται η ψηφορία. Λήξη. Τερπολογία 5317 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε στην 5318. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 5319. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 53-20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53-21. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται 53-22 άρχεται η ψηφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 53-23 Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο. Τροπολογία 53, 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παρακαλώ. Ο κ. Δικάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξηγήσω τη φύση της 5345 που έχει κατατεθεί από μένα και να την εξηγήσω κυρίω στον εισηγητή, στον κύριο Γιάρη και ελπίζω την υποστηρίξει. Πρόκειται για μια τροπολογία που δημιουργεί τις συνθήκες για ένα ταμείο αναδιάρθρωσης ε, κατόπιν ε, της λήξης ε, των επιδοτήσεων για τη ζάχαρη το 2017. Ξέρετε τι έγινε με την πολιτική της ζάχαρης το 2007, έτσι ανάλογα όλα τα εργοστάσια που θα πρέπει να κλείσουν ε, στην Ευρώπη στο μέλλον πρέπει να έχουν το δικαίωμα για να μπορούν να διατηρήσουν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πνεύμα ε, της τροπολογίας που έχω καταθέσει και ελπίζω να τη δεχτούν οι περισσότεροι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Μήπως ε, να μας πείτε πιστεύει και ο ε, Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Ντεκάστρο που διευκρίνησε ότι πρόκειται για δύο θέματα. Το ένα είναι τα καθαρά νούμερα και το άλλο είναι το πολιτικό μήνυμα και υπ' αυτή την έννοια του πολιτικού μηνύματος συστήνω να με την τροπολογία αυτή. Νομίζω ότι είναι καλό το μήνυμα που θα προέλθει από την Επιτροπή αυτή. Λέω λοιπόν να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της τροπολογίας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σίγητη. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία για την 5345 κατόπιν ε, της προφορικής ε, παρουσίασης της τροπολογίας του κ. Ντεκάστρο. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία του κ. Ντεκάστρο 5345. Πέρας. Α, δεν είχα πει ότι υπήρχε λήξη της ψηφοφορίας, συγγνώμη. Τώρα, λίγουμε την ψηφοφορία εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κύριε Σιγητά. Περνάμε τώρα στην 5347. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 5347. Ευχαριστώ, πέρας. Απορρίπτεται. Κατόπιν περνάμε στην 5349. Άρχεται η ψηφοφορία. 5349. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 5350. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 53-51. Άρχεται η ψηφοφορία για την 53-51. Ευχαριστώ. Πέρας. Πέρας. Ψήφισατε όλοι. Ωραία, εγκρίνεται. Περνάμε στην 53-52. Άρχεται η ψηφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Κατόπιν περνάμε στην 53-53. Άρχεται ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5360, άρχεται η ψηφοφορία για την 5360. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα τροπολογία 53-54 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53-56. Άρχεται η ψηφοφορία για την 53-56. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 53-58. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 53-59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53-63. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Λήξη. Απορρίπτεται. 53-64. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53-65. Άρχεται η ψηφοφορία. απόφαση. Απορρίπτεται. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Για το σχέδιο γνωμοδότησης. Το διορθωμένο. Δεν ξέρω αν ε, θέλετε το λόγο κύριε Σιγητά. Λοιπόν, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Ο συλλογητή δεν θέλει να πει κάτι. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. καρας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Τροπολογία 11. Τροπολογία 11 παρακαλώ. Διόρθωση. Όχι. Την 5 θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 8. Ευχαριστώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 7. 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 11. 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 10. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 12. 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 13. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορριφθήκε. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 14. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 15. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 15. Εύχομαι να μην ψηφίσω, απλώς να σας ε, υπενθυμίσω την τροπολογία μου. Όπως σας είχα ζητήσει, προτείνω μια προφορική τροπολογία που τροποποιεί την ε, τροπολογία που είχα αποβάλει, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προσέξουν ιδιαίτερα τον τομέα του ρυζιού και να επισημάνω την σημασία της προστασίας των καταναλωτών από τις εισαγωγέ ε, ρυζιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο τομέας ε, του ε, ρυζιού, κυρίως του ιταλικού ρυζιού, είναι ένας τομέας υψηλής ποιότητας, ο οποίος θα πρέπει κατά την άποψή μου να προστατεύεται και ενώπιον των εργαζομένων, εργαζομένων και σε άλλες χώρες του κόσμου, οι οποίοι εργάζονται σε συνθήκες μεσαίωνα και επομένως είναι αθέμητος αυτός ο ανταγωνισμός, διότι οι τιμές παραγωγής για το ρύζι είναι τελείως διαφορετικές, ε, δεδομένου ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές εργασιακές συνθήκες. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την Επιτροπή και από τον εισηγητή να δεχτούν ε, την ε, τροπολογία για να μπορέσουμε να δώσουμε και ένα ε, μήνυμα στους ε, παραγωγούς ε, ρυζιού και να ευχαριστήσω και τον κύριο Ταραμπέλα που μου έδωσε συμβουλές για το πώς πρέπει να κάνω την τροπολογία. Τον αγαπώ πολύ γιατί εγώ είμαι μικρός και δεν ξέρω. Ας μην ε, ξαναγυρίσουμε στο θέμα του κυρίου Τάραμπέλα. Ο κύριος Άγνιου ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, σωστά κατάλαβα ότι επρόκειτο για προφορική τροπολογία. Γιατί αν, είναι, αν πρόκειται περί προφορικής, εγώ είμαι κατά, όχι ως προς την ουσία, αλλά Ξέρετε ότι αυτό το κάνω ως θέμα αρχή, το ήξερε και ο προηγούμενος πρόεδρος. Πρώτον, το ανεξάρτητο κόμμα της Αγγλίας ε, έχει ως σκοπό να μην βοηθάει το θεσμικό αυτό όργανο και επίσης αυτή η συνήθεια των προφορικών τροπολογιών μπορεί να γίνει μεταδοτική και μπορεί να οδηγήσει σε κακή νομοθεσία και θα ξέρετε ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένο στην Ολομέλεια ο οποίος ε, κάνει μακροσκελείς ε, προφορικές τροπολογίες που κανείς δεν καταλαβαίνει. Η μόνη εξαίρεση στο γενικό κανόνα είναι για λόγους ευγενία στους δύο συναδέλφους στην ομάδα EFD. Είμαι, ε, δεν είμαι καθόλου δημοφιλής αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μου να γίνω δημοφιλής. Αν ε, ξέρετε ε, πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι και ένας να, αν υπάρχουν το προφορικές τροπολογίες είναι καταδικασμένες γιατί είμαι εγώ εδώ και ένας να έχει αντίρρηση καταπίπτει. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν ένσταση εδώ, αντίρρηση. Πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε για το αν πρέπει να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία και μετά θα ψηφίσω με την ίδια την τροπολογία. Πρώτα λοιπόν ψηφίζομαι με εξή αντικείμενο. Θα την ψηφίσω με αυτή την τροπολογία ή όχι. Δηλαδή είναι, είναι παραδεκτή. Αυτό θα ψηφίσουμε πρώτα. Αν κρίνουμε παραδεκτή την τροπολογία αυτή για να την ψηφίσουμε. Αυτό μου λέει η γραμματεία. Ο κύριος Γιάρ. Κύριε Πρόεδρε, τη διαδικασία, στη διαδικασία δεν είμαι τόσο άκαμπτος όπως εσείς, αλλά αν θυμάμαι καλά η προφορική τροπολογία μπορεί να ε, γίνει ε, αποδεκτή αν δεν ψηφίσει κανείς κατά. Δηλαδή ο συνάδελφος έχει δίκιο που είπε ότι αφού είναι κατά η προφορική τροπολογία δεν τίθεται καν, δεν υφίσταται. Επειδή έχει, ε, ε, υποβάλλεται καθυστερημένα, θα πρέπει να ξεπεράσει πολύ περισσότερα εμπόδια από τη μια ε, κανονική τροπολογία. Ναι, ίσως ο επικεφαλής της γραμματείας μου θα μας το εξηγήσει. Αν 10% των μελών έχουν ένσταση σε προφορική τροπολογία δεν μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία. Αυτό σημαίνει δύο μέλη τουλάχιστον, δύο μέλη τουλάχιστον από αυτή την Επιτροπή. Δύο πρέπει να έχουν ένσταση. Τότε δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία. Χρειάζονται δύο. Ο κύριος Σάγνου είναι ένας. Αν υποστηρίζει και κάποιος άλλος, αυτομάτως καταπίπτει η προφορική τροπολογία. Ο κύριος Ταραμπέλα. Είπατε ότι χρειαζόμαστε 10% των μαλλών. 10% ε, είναι 4 ή 5 στους 42, επομένως δεν είναι 2. Θα ήθελα να σας προτείνω το εξής λοιπόν εάν συμφωνεί και ο Πρόεδρος, να κάνουμε μια επαλήθευση για να είμαστε απόλυτα βέβαιοι και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σημεία της ε, ψηφοφορίας και να επανέλθουμε στο σημείο αυτό στο τέλος για την προφορική τροπολογία και την ε, τροπολογία και τη διαδικασία. Εντάξει, θα το εξετάσουμε. και θα δούμε πώς θα χειριστούμε την ένσταση του κυρίου Άγνιου. Νομίζω ότι ζητεί το λόγο. Παρακαλώ κύριε Άγνιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με, με ενδιαφέρον βλέπω ότι δημιούργησε μια δυσφορία όλο αυτό, αλλά στην προηγούμενη θητεία ένας χρειαζόταν για να καταπέσει. Ο προηγούμενος πρόεδρος το είχε δεχτεί αυτό. Αν δεν υπάρχει αλλαγή στους κανονισμούς και αν δεν έκανε λάθος ο προηγούμενος πρόεδρος, ε, Έχουμε πρόβλημα εδώ. Νομίζω ο προηγούμενος πρόεδρος είχε δίκιο. Α, όντως ε, ε, αυτοί ήταν οι κανόνες. Εν τω μεταξύ μπορεί να άλλαξαν. Θα ζητήσω να το ελέγξει αυτό η γραμματεία για να είμαστε απόλυτα βέβαιοι σχετικά με τον αριθμό των απαιτουμένων ενστάσεων. Αν είναι ένας που χρειάζεται ή το 10%. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη γραμματεία πάνω σε αυτό. Οπότε ας περιμένουμε, αφήνουμε στην άκρη αυτή την τροπολογία και προχωρούμε στην τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ευχαριστώ. Δεκτή. Προχωρούμε στην 21. Όχι. Συγγνώμη, την 22, γιατί η 21 έχει αποσυρθεί. 22 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία της 22. Ευχαριστώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. Προχωρούμε. Τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι η τροπολογία του κυρίου Ταραμπέλα. Ευχαριστώ. Πέρας. εγκρίνεται. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε πώς θα χειριστούμε το θέμα που απομένει. μας εξηγήσει η Γραμματεία. Υπάρχει ο αλλαγή στον κανονισμό. Ο κανόνας που εφαρμόζεται είναι ότι στην Ολομέλεια 40 μέλη μπορεί να είναι κατά ε, μιας προφορικής τροπολογίας και ένα αντίστοιχο ποσοστό μπορεί να εφαρμόζεται στι ε, επιτροπές και επομένως ε, για τα 40 η αντιστοιχεία είναι τρία μέλη στην Επιτροπή Γεωργίας. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν τρεις ενστάσεις για την προφορική τροπολογία ώστε να μην μπορέσει να ε, ψηφιστεί. 169 το άρθρο το σχετικό του κανονισμού. Χρειαζόμαστε τρία μέλη. Ο κύριος Άκνιου είναι κατά. Εάν υπάρχουν άλλα δύο μέλη τα οποία είναι, ε, τάσσονται υπέρ του κυρίου Άγνου, τότε δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία του κυρίου Μπονάνου. Λοιπόν, με βάση αυτή την εξήγηση ρωτώ, υπάρχουν άλλοι που ενίστανται, όπως και ο κύριος Άγνιου. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Μπονάνο πρέπει να επαναλάβει την τροπολογία του. Υπάρχει και άλλη ένσταση. Πείτε μας. στην Ιρλανδία. Μια ένστασή μου κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι οι πολιτε δεν καταλαβαίνουν τι πολυπλοκότητε και τους κανόνε. Και έρχομαι εδώ και ανακαλύπτω ότι ούτε και η γραμματεία δεν καταλαβαίνει τις, τους κανόνες. Οπότε τι στο καλό ε, δυνατότητα έχουν οι απλοί πολίτες. Ο κύριος Νίκολσον επαναλαμβάνω ότι η γραμματεία ε, έχει δίκιο. Αυτό που είπε η γραμματεία απεδείχθη αληθινό, γιατί οι κανόνες εδώ μεταξύ άλλαξαν. Ο κύριος Νίκολσον. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι κάνουμε στο γόνατο τους κανόνες. Δεν έχω πιστεί 100% από αυτά που άκουσα. Επειδή είναι κανονισμός στην Ολομέλεια, δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά ισχύει και στην Επιτροπή αυτό. Θέλω αυτό να πάει στην Επιτροπή Κανονισμού του Κοινοβουλίου για να ελεγχθεί και πάλι, γιατί εγώ άλλα είχα υπόψη μου και με κάθε σέβας, εγώ δεν ε, θεωρώ ότι είμαι ειδικό για τους ε, κανόνες, αλλά δεν είναι ωραίο να καθόμαστε εδώ και να μην ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι ο κανονισμός. Εμείς φαίνεται ότι δεν είμαστε βέβαιοι σχετικά με τους δύο ή τους τρεις. Νομίζω μπορεί να έχει δίκιο ο κύριος Άγνιου. Α, εγώ μπορώ να είμαι ο δεύτερος που έχω ένσταση. Αν υπάρξει και ένας τρίτος μπορεί να μην περάσει η προφορική τροπολογία. Παρακαλώ, χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά είναι πονίδιστο αυτό το γεγονό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν, πεθαίνουν από την πείνα, υπάρχουν προβλήματα εμπορίου, προβλήματα γεωργών που δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους και εμείς καθόμαστε εδώ με 5.000 ε, γραφειοκράτου ε, ε, γραφειοκράτους ε, να συζητάμε για το αν ισχύει μία ψήφο ή δύο ψήφοι, δεν, μπορούμε δεν ξέρουν τι του γίνεται. πραγματικά είναι ντροπή. Ο κύριος Φλάνναγκαν. προτάθηκε ότι δεν έχει πρόβλημα με τη γραμματεία γιατί είχε δίκιο. Είναι άλλο να μαντεύεις αν έχεις δίκιο και τελικώς να έχεις δίκιο και άλλο να έχεις δίκιο. Ε, επαναλαμβάνω ότι απλώς με επίθετε για αυτό που σας είπα προηγουμένως ε, πριν έρθω εδώ. Όλα αυτά είναι ένα τσίρκο εδώ μέσα. Κύριε Σιγητά. Τελευταία παρέμβαση παρακαλώ. Ο κύριο Γιάρ. Äh, ε, θα έλεγα μετά τη συζήτηση ότι συμφωνώ με τον συνάδελφο να μην ε, ψηφιστεί η τροπολογία, να προσθέσω και εγώ το όνομά μου δηλαδή και να διευκρινίσουμε το θέμα για να ξέρουμε πότε γίνεται ε, παραδεκτή ή όχι μια προφορική τροπολογία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ο δεύτερος. Αν υπάρξει και τρίτος, τότε τελειώνει το θέμα. Νομίζω ότι οι προφορικές τροπολογίες πρέπει να είναι η εξαίρεση και το ξέρουμε. Κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να μελετά καλά τις τροπολογίες, αυτό δεν γίνεται στις προφορικές. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί, γιατί όταν έχουμε προφορικές τροπολογίες ε, θα πρέπει αμέσως να μπούμε στο νόημα. Ε, τρεις, ε, μπορώ να προσθέσω και εγώ το όνομά μου, άρα υπάρχει να υπάρξει και ένας τρίτος. Ωραία. Ήταν και ο κύριος Νίκολσον κατά της τροπολογίας και όπως και ο κύριος Άγνου, τώρα και ο κύριος Γιάρ, επομένως έχουμε τρεις κατά της προφορικής τροπολογίας, επομένως δεν θα ψηφιστεί αυτή η προφορική τροπολογία. Θα ήθελα να ζητήσω βέβαια από τη Γραμματεία της Επιτροπής να θέσει το ερώτημα στην Επιτροπή Κανονισμού. Και θεωρώ ότι κάποια από τα σχόλια τα οποία έγιναν εδώ είναι μάλλον υπερβολικά. Σε αυτή την περίπτωση η γραμματεία έχει δίκιο και θα δώσω το λόγο στον επικεφαλής της γραμματείας αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να σας ε, ε, πω ότι όντως έγινε αλλαγή του κανονισμού. Στο παρελθόν ένας βουλευτής αρκούσε να υποβάλει ένσταση για να μην γίνει αποδεκτή μια προφορική τροπολογία προς ψήφιση. Τώρα ο κανονισμός προβλέπει ότι στην Ολομέλεια θα πρέπει να είναι 40 τα μέλη τα οποία θα πρέπει να ενίστανται για να μην ληφθεί υπόψη μια προφορική τροπολογία και επειδή για πρόκειται για έναν κανονισμό της Ολομέλειας ο οποίος ισχύει μουτάτης μουτάντης και στις αρμόδιες επιτροπές ε, λαμβάνουμε ότι θα πρέπει αντιστοίχως, κατά αντιστοιχεία λοιπόν, να έχουμε τρία μέλη ε, της Επιτροπής, ε, τα οποία να ενίστανται για να μην γίνει δεκτή μια τροπολογία. Ε, επιβεβαιώνω ότι έγινε αλλαγή του κανονισμού και δεν είναι η γραμματεία αυτή η οποία άλλαξε τον κανονισμό. Σημειώνουμε λοιπόν αυτές τις πληροφορίες και θα ήθελα να ζητήσω να μας τα δώσετε και γραπτό όλα αυτά, ώστε στο μέλλον να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους νέους κανόνες ε, του κανονισμού. Ο κύριος Άκνου καταρχάς. Παρακαλώ. να κάνω κάποια σύντομα συμπεράσματα. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι που κατάφερα ε, η Βόρεια Ιρλανδία και η Νότια Ιρλανδία να συμφωνήσουν για κάτι. Και δεύτερον, υπάρχει ε, πιθανότητα τα όσα έκανα εγώ στην προηγούμενη θητεία να υποχρέωσαν το Κοινοβούλιο να αλλάξει τους κανόνες. Σας ευχαριστώ. E, ε, ουδέν σχόλιο. Παρακαλώ κύριε Μπονάνο. Ειλικρινά με εκπλήσει που είναι μέλος του κόμματος του Φάραντς είναι τόσο περήφανος που κατάφερε να ε, παρακολύσει μία ε, ψηφοφορία. Είστε μεν αντιευρωπαϊστής, αλλά πραγματικά ε, εδώ πέρα τι κάνετε για να πειράξετε τη γυναίκα σας. Αφαιρείτε μέλη του σώματός σας. Τι να σας πω, εγώ είμαι δήμαρχος μια μικρής Ιταλικής πόλης, ο οποίος ήρθε εδώ με πολύ μεγάλη ελπίδα ώστε να προσπαθήσει να ε, επιτύχει μια Ευρώπη που να είναι πολύ πιο κοντά στους πολίτες. Πραγματικά ε, οι γεωργοί ε, πίστευαν ότι θα μπορούσαν για παράδειγμα να αλλάξουν ένα πολύ μικρό κανένα. Πραγματικά οι γεωργοί χρειάζονται απαντήσεις και όχι η γραφειοκρατία η οποία είναι αυτή η οποία οδηγεί στο θάνατο αυτή την Ευρώπη. Πραγματικά ντρέπομαι που άκουσα συγκεκριμένα πράγματα γιατί εγώ δεν έχω έρθει εδώ για να παίξω. Προσπαθώ να επιτύχω κάποιο αποτέλεσμα για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε αυτό το τομέα. Και εμείς τι κάνουμε, καθόμαστε εδώ και συζητάμε αν χρειαζόμαστε μία ψήφο ή τρεις ψήφους και αυτοί γελάνε για αυτά που πρέπει να γίνουν. Πραγματικά θα έπρεπε να ντρέπονται. Πρόκειται για το καρκίνωμα της Ευρώπης. Είναι σαφές αυτό. Είναι το καρκίνωμα της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να υπερασπιστεί κάποιο τη Γεωργία με αυτόν τον τρόπο. Δεν την υπερασπιζόμαστε έτσι. Θα το πω εδώ, θα το πω και έξω και πραγματικά θα έπρεπε να του πάρει κάποιο με τις κλωτσιές γιατί θα έπρεπε να ντρέπονται για αυτά που λένε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα σας παρακαλώ να σας ζητήσω να μην υπερβάλλουμε τόσο ε, με σχόλια που δεν είναι καθόλου πολιτικά χαρακτήρα. Αυτά είναι τα πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι έχουν οι κανόνες και Δυστυχώς ε, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την τροπολογία με αυτόν τον τρόπο. Λυπάμαι που δημιουργήθηκε αυτή η σύγχυση, αλλά όπως μας είπε και η γραμματεία, άλλαξαν οι κανόνες και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουμε. Να περάσουμε στη συνέχεια στο ε, ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Γνωρίζω ότι ο καθής έχει δικαίωμα στην απόψη του, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει και αυτό το ρόλο του να διαδραματίσει. Να περάσουμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 7 για την υγεία των ζώων. Επιβεβαίωση της θέσης σε πρώτη ανάγνωση και ορισμός της διαπραγματευτικής ομάδας. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε επισήμως για τη διαδικασία της συναπόφασης. μετά την ανάλυση που έγινε και την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νομοθεσία για την υγεία των ζώων, ε, τη οποία εισηγήτρια είναι η κυρία Πόλσεν, και ε, τα προστατευτικά μέτρα ε, φυτοϊγείας συζητήθηκαν και η Ευρώπη των Συντηρητικών και ε, Δημοκρατών χρειάζεται να ορίσει νέο εισηγητή για τη δεύτερη ανάγνωση. Η Επιτροπή ε, αποφάσισε σχετικά για την ανανέωση της ε, διαδικασίας με βάση την πρώτη ανάγνωση η οποία εγκρίθηκε στις 15 Απριλίου του 2014. Βάσει του άρθρου 73 η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει επίσημη απόφαση όσον αφορά το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων επί τη βάση αυτής της συγκεκριμένη εντολής και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδος. Θα ήθελα λοιπόν να ψηφίσουμε αυτές τις αποφάσεις, καταρχάς όσον αφορά τη διαδικασία για την υγεία των ζώων και ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έχουμε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες. Πρώτη ψηφοφορία για την ε, ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων μετά την επιβεβαίωση της θέσης μας σε πρώτη ανάγνωση. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για αυτό το πρώτο σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα της ψηφοφορίας. Κατόπιν. Ψηφοφορία για, την, ε, για τον ορισμό της διαπραγματευτικής ομάδας και για τον εισηγητή και για τους κοιόδες εισηγητές. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρασε τη ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη συνέχεια στο σημείο 8. Αγροφάγκο προστατευτικά μέτρα για ε, τα επιβλαβή ε, για, τα φυτά το, για τα φυτά οργανισμούς για τους επιβλαβείς συγγνώμη, για τα φυτά οργανισμούς. Και πάλι εδώ θα πρέπει να ε, ψηφίσουμε για την ε, συνέχεια ε, της επιβεβαίωσης της θέσης πρώτη ανάγνωση και, για τον ορισμό της διαπραγματευτικής ομάδας. Και πάλι ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιβεβαιώσει λοιπόν αν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις εν ώψη μιας δεύτερης ανάγνωσης ε, λόγω της θέσης μας σε πρώτη ανάγνωση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η τροπολογία η διαδικασία ε, και τώρα περνάμε στον ορισμό της διαπραγματευτικής ομάδας. Έχουμε πρόεδρο, εισηγητή και σκιώδης εισηγητής και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρασε της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Και στη συνέχεια, σημείο 9. Σημείο 9. Ζωοτεχνική και γενολογική όρη που εφαρμόζονται στο εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση Ζώνων Παραγωγής και των απαραγωγικού υλικού τους. Ο στόχος είναι να προωθηθεί το ελεύθερο εμπόριο αυτών των ζώων και του γενετικού του υλικού, του αναπαραγικού του υλικού, έχοντας κατά νου και τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων και τη συντήρηση των γενετικών πόρων. Το σχέδιο κανονισμού περιλαμβάνει διάφορες πτυχές της νομοθεσίας της ζωοτεχνικής σε ένα ενίο νομικό πλαίσιο και προσφέρει και μία νομική βάση για την έγκριση των εξουσιοδότηση πράξεων και των ε, εκπαιδευτικών μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο, στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας παρουσιάσουν τα κυρία στοιχεία της πρότασης. Έχετε το λόγο. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος θα πάρει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω ένθερμα. Και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να παρουσιάσω το σημείο. Καλημέρα σας, λέγομαι Μάιλερ της Λαυμίσκο και προέρχομαι εγώ τη γαμάδα. Δέλτα Σάνκο, είμαι πληρωτής Γενικός Διευθυντής. Να ξεκινήσω με μία σύντομη εισαγωγή των ε, λόγων και των ε, στόχων αυτής της πρότασης. Όπως μπορεί να γνωρίζετε, σήμερα η ζωοτεχνική νομοθεσία στην Ένωση αποτελείται από τέσσερες ε, βασικές ε, πράξεις ε, οριζόντιες που παρουσιάζουν κάποια μέτρα για την έγκριση και την καταλογοποίηση των επιχειρήσεων και επίσης και την καταγραφή των ζώων σε διάφορα είδη μητρώων. Ε, οι κανόνες και η γενετική αξιολόγηση και το περιεχόμενο των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών ε, για τα ζώα ε, εκμετάλλευσης και τα ζώα εκτροφής. Έχουμε διάφορες οδηγίες που έχουν εφαρμοστεί με κάπως διαφοροποιημένους τρόπους στα κράτη-μέλη και αυτό έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα στο εμπόριο, στον στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα φυσικά υποχρεωθήκαμε να λησαυνοποιήσουμε αυτό το δήμα της νομοθεσίας. Έτσι λοιπόν ο κύριος στόχος του προτινόμενου κανονισμού ε, για τους ζωοτεχνικούς όρους βασίζεται στα άρθρα 42 και 43-2 της συνθήκης για την ενοποίηση των τεσσάρων ε, οδηγιών σε έναν κανονισμό που να καλύπτει όλο το ζωοτεχνικό και εκτιμένο σε ό,τι αφορά τα σημαντικά οικονομικά είδη ή τα είδη που είναι σημαντικά για το εμπόριο από τη σκοπιά του αναπαραγωγικού υλικού και ποιος έχουμε και διατάξεις για επίσημους ελέγχους που σήμερα υπάρχουν σε οδηγίες για κτηνιατρικούς ελέγχους και για σε συνεργασία με τις αρχές που θα καταργηθούν όταν τη στιγμή αυτή τη στιγμή που θα το κείμενο του νέου κανονισμού. Έτσι λοιπόν, αν υιοθετηθεί ο νέος κανονισμός θα έχουμε ασφάλεια δικαίου και αποσαφήνιση του θέματος των επίσημων ελέγχων. Έτσι θα έρθουν ε, τα ε, εμπόδια που έχουν παρατηρηθεί στο εμπόριο και ορισμένα κράτη-μέλη έχουν καταγγείλει ότι υπάρχουν ε, τέτοια εμπόδια και σε ορισμένες ε, περιπτώσεις ε, υπήρξε πρόβλημα με την εγκατάσταση κάποιων ε, εταιριών που είχαν εγκριθεί σε άλλα κράτη-μέλη. Η εισαγωγή, μάλλον υπάρχει, υπάρχει τώρα μία διαφορά γιατί γενικά φύγονται όλα τα είδη των ζώων, όμω, η νέα πρόταση ενδυναμώνει την υιοθέτηση των κατεξιζώτης πράξεων για, ε, για την αναπαραγωγή καθαράς φυλής και άλλων ζώων, αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τη λειτουργία τη εσωτερικής αγοράς ή για το προστατευμένο αναπαραγωγικό υλικό. Η πρόταση βασίζεται σε εφιστάμενη νομοθεσία στο ζωοτεχνικό τομέα, αλλά και στη νέα πρόταση για τους επίσημους ενέχους και στις ευρύς συζητήσει που υλοποιήθηκαν στη μόνιμη επιτροπή για τους ζωοτεχνικούς όρους και επί συγκεκριμένων δραστηριοτήτων διασυνοριακού χαρακτήρα των εταιριών εκτροφής και επίσης ε, λάβουμε υπόψη και διάφορες καταγγελίες από τις εταιρείε και από τις εκτροφείς και επίσης ε, ζητήθηκαν και διευκρινήσεις από τις αρμόδιες αρχές και από συγκεκριμένα κράτη-μέλη, κυρίως ε, για το θέμα της εκτροφής των αλόγων. Με αυτή λοιπόν την πολύ σύντομη εισαγωγή. Ελπίζω ότι θα μπορούσατε να μας υποστηρίξετε για αυτή την ε, προτινόμενη ενοποίηση σε ένα κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε στη συζήτηση. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση. Πιστεύω ότι ε, αυτή η δήλωση απλούστευσης, δηλαδή ότι σε ένα κείμενο θα ενοποιήσουμε διάφορα ισχύοντα κείμενα, είναι κάτι θετικό. Αλλά αν δούμε την πρόταση λεπτομερώς, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε το σύνολο των ειδών και των φυλών και τελικά καταλήγουμε σε μία μέγιστη πολυπλοκότητα των διατάξεων και για το τι θα πρέπει να κάνουν οι φορείς και εγώ κατάλαβα ότι διακυβεύονται πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την εκτροφή αλόγων όμως καταλαβαίνω γιατί θα επιβάλλουμε τις ίδιες συνθήκες ε, σε όλα τα είδη. Ε, η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που, συζητούνται, που από αυτό το κείμενο είναι εκτός εμβέλειας ε, για ορισμένους επιχειρηματίες. Αν ε, η Κομισιόν ε, θέλει ε, να αναφερθεί σε συγκεκριμένες φυλές ράτσες που είναι σημαντικές, νομίζω ότι πρέπει να το πει σαφώς γιατί τελικά θα καταλήξουμε στο απλώς να διατηρήσουμε κάποιες μεγάλες ράτσες φυλές στην Ευρώπη. Επίσης διαπιστώνουμε εκτός κι αν είμαι κακός πληροφορημένος, ότι δεν έχουμε ακόμη μάθει τι έγινε με τη μελέτη αντικτύπου για το κείμενο αυτό. Και αν υπήρξε μελέτη αντικτύπου, καλό θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω ο εισηγητής της Επιτροπής μας και της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, να λάβουν αυτή την μελέτη αντικτύπου. Εγώ τέλος πάντων ε, είμαι ε, εισηγητής μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και μπορώ να πω ότι θα είμαι και αρνητικός απέναντι σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βαλκάψελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η θέση της Ισπανίας ε, επίσης είναι επικριτική για διάφορες ε, πτυχές ε, της πρότασης της Κομισιόν. Αφενός, ε, κατανοούμε ότι εδώ επικεντρωνόμαστε στις ανταλλαγές που γίνονται από ιδιώτες και επιχειρήσεις πολυεθνικές πολλές φορές. Όμως είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ειδική μεταχείριση για τις αυτόχθονες φυλές που κινδυνεύουν από εξαφάνιση και μπορούν να αποτελούν οικονομική δύναμη. Από την άλλη, προτείνει ο οικονομισμό την απελευθέρωση των προγραμμάτων βελτίωση. Όμω, ε, αυτή η απελευθέρωση, αν δεν γίνει με ομοιογενέ τρόπο, αυτά τα προγράμματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια απώλεια τη ποιότητα των φυλών. Και επίση, ε, ε, ε, ότι οι έλεγχοι στις εμπορικές ανταλλαγές, όμως θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι και στις ενώσεις των κτηνοτρόφων και στους ίδιους τους εκτροφείς. Σε αυτή την νομοθεσία εμπλέκονται τα υβριδικά, υβριδικές φυλές όπως παραδείγματος χάρη η χείρη, η υβριδική χείρη με τις καθαρές φυλές. Εδώ πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο κανονισμός θα έπρεπε να τα αποσαφηνίσει αυτά με σαφήνεια ή θα έπρεπε να υπάρχουν ξεχωριστά νομοθετήματα. Επίσης, κατανοούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπαίνει υπερβολικά σε νομικά θέματα όπως η άδεια, ε, οι ονομασίες σε θέματα εκτροφών και νομίζω ότι αυτά είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας, επομένως δεν σέβεται εδώ η Επιτροπή την αρχή της επικουρικότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φέραντ. Ναι κύριε Πρόεδρε, όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ε, τα δει όλα. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ε, ταρτάρα από κρέα αρολές. Ε, σας καλώ να το κάνετε στη Βουργουνδία σε επόμενε διακοπέ Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ αποδυναμωμένο το κείμενο και δεν προστατεύει τις δυνατότητες εκτροφής αρκετά. Αν δούμε τη γαλλική περίπτωση για παράδειγμα, εμείς έχουμε περίπου 40 ε, διαφορετικές ε, ράτσες. Πρόκειται για πολιτιστική κληρονομιά ε, την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε και αυτή θα πρέπει να σχετίζεται και με τον τόπο καταγωγής. Πρόκειται για οικονομικό ε, όφελος, διότι πολλές από αυτές τις ράτσες είναι παγκοσμίως γνωστός και επομένως αυτό αποτελεί ε, όφελος για τη χώρα μας. Δεν προστατεύονται λοιπόν επαρκώ οι χώρες που έχουν ένομα δικαιώματα και πραγματικά ε, οι ράτσε αυτέ αποτελούν τμήμα τη ιστορία του ε, και του τόπου του. Για παράδειγμα η κατηγορία Σαρολέ θα έπρεπε να παραμείνει και δεν θα πρέπει ε, κάποιοι να οικειοποιηθούν τη γενετική τους ποιότητα. Όπως γίνεται λοιπόν και με τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα, αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να προστατεύσει κάποιος τον τόπο και την κληρονομιά του. Ähm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά τους προλαλήσαντες συναδέλφους θα είμαι συντομότατος. Νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το κείμενο ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει στις μικρές κυρίως βόηες φυλές γιατί θα ήταν αρκετά παράλογο να δώσουμε ένα σωρό λεφτά για αυτές τις ε, βόηες ε, απειλούμενες από εξαφάνιση φυλές, να τις προφυλάξουμε ή να τις ε, προστατεύσουμε και από την άλλη να δυσκολεύουμε με τους κανόνες μας τη ζωή των εκτροφέων. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε πολύ προσεκτικά όλα αυτά και να δώσουμε μηνύματα ότι οι εκτροφείς δεν θα δουν να δυσκολεύεται το έργο τους ε, μέσα από τους κανόνες για τις φυλές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα άμεσο ερώτημα. Εδώ θέλουμε να νοικοκυρέψουμε απλώς ε, τους κανονισμούς μας ή αποσκοπούμε και στην πιθανή εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες όπου προετοιμαζόμαστε για τις συζητήσεις αυτές και θέλουμε όλα να είναι διευκρινισμένα και ε, ενοποιημένα σε ένα κείμενο. Οι απλές ερωτήσεις είναι οι δυσκολότερες και ο παρακαθήμενος βουλευτής Υπάρχουν ε, συγκεκριμένα είδη τα οποία πρέπει να προστατευτούν, αυτόχθονα είδη, βοηδή. Για παράδειγμα, εμείς ε, προσπαθούμε να προστατεύσουμε ένα συγκεκριμένο είδο της ίστρια, το οποίο ήταν αυτόχθονο στην περιοχή. Ε, ξοδέψαμε πάρα πολλά χρώματα και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και όλα αυτά αυτή τη στιγμή αντιστρέφονται. Γι' αυτό ακριβώ και υποστηρίζω πλήρω ε, την ευρωπαϊκή κληρονομιά, ιδίως όταν πρόκειται για συγκεκριμένε ράτσες και είδη, η Κροατία, η Ιταλία, ε, η Ισπανία έχουν πάρα πολλά αυτόχθονα είδη και αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν ε, ετοιμάζουμε κάποιο συγκεκριμένο κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάκοβιτς ήταν ο μιλητής που ακούσαμε μόλις τώρα. Και τώρα η κυρία Σενέα. Για να... εγώ είμαι υπέρ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θέλω να πω, και μην βάζουμε σε κίνδυνο τι αυτόχθονε ράτσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στη Γαλλικία, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την παραγωγή βόλου κρέατος, του χάρη. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα έτσι όπως παρουσιάστηκε η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Και ένας ακόμη ομιλητής, κυρία Μόρι. Και εγώ είμαι αντίθετη σε αυτό το αίτημα. Νομίζω ότι θέτει σε κίνδυνο τις αυτόχθονες ε, ράτσες ε, υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στην Ιταλία και στη Ισπανία και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι έγινε και με τους σπόρους και με την βιοπικιλότητα. Στο μέλλον θα διευκολυνθούν οι πολυεθνικές να μπορούν να καταγράφουν αποκλειστικά το γονιδίωμα των ζώων. Γι' αυτό λοιπόν είμαι κατά της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Ευχαριστώ όλους για τις απόψεις και ερωτήσεις. Και τώρα ο κύριος Μίκο από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ θα απαντήσει. Θα, θα, και θα εξετάσει τα θέματα. Αξιότιμα μέλη, επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι στην προσπάθεια τις διατάξεις τεσσάρων οδηγιών να τις εντάξουμε σε ένα κανονισμό δεν ε, πιάσαμε μια βασική αρχή όπως λειτουργεί σήμερα. Δεν υπάρχει αλλαγή αρχή στην προσέγγιση ε, σε κανένα κείμενο. Αν πρόκειται για κάποια αλλαγή, έχουμε μια ελαφρά αυξημένη προστασία ε, στις ε, μικρές βόλες φυλές. Ε, η πρόταση παραμένει ως είχε στον προηγούμενο κανονισμό. Τώρα, σχετικά με τα σχόλια που αφορούν την υψηλότερη πολυπλοκότητα της ε, πρότασης πρέπει να εξηγήσω ότι παλιότερα είχαμε τέσσερις οδηγίες οι οποίες όμως εφαρμόζονταν με διαφορετικούς τρόπους στα κράτη-μέλη στην πραγματικότητα. Τώρα η περιπλοκότητα είναι πολύ ε, ε, μεγάλη και υπήρχαν διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη-μέλη. Τώρα έχουμε ένα κείμενο σαφές, συνεκτικό, εφαρμοστέω σε όλα τα κράτη-μέλη με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που θα διευκρινίζει τα πάντα και τις αλλαγές κατανόησης του παρόντος πλαισίου. Μπορεί να έχουμε περισσότερο κείμενο, αλλά είναι απλούστερο στην πραγματικότητα και ισχύει το ίδιο σε κάθε κράτος μέλος. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, προστιθέμενη αξία της πρότασης που αντανακλά και, και καλύπτει και πολλά παράπονα που είχαμε ακούσει σχετικά με τη διαφορετική κατανόηση και νομική ε, εξήγηση στα κράτη-μέλη. Τώρα, ε, γιατί ε, το απλό ερώτημα που ακούσαμε έχω και από εγώ απλή απάντηση. Καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις με τις ΙΠΑ τη Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου. Έχει να κάνει μόνο με τις προσπάθειες που κάναμε και την προηγούμενη περίοδο και αυτό τεκμηριώνεται. Προσπάθειες απλούστευσης του κεκτημένου στην υγεία των ζώων και στους συναφείς τομείς ε, των τροφίμων γιατί υπήρξαν εξελίξεις μακρές ε, περισσότερο μακρές από τις άλλους τομείς. Είχαμε αρχίσει πριν από 40-50 χρόνια τις υποθέσεις αυτές και έπρεπε να εξυγχρονίσουμε. Έπρεπε λοιπόν να ενοποιήσουμε, να βοηθήσουμε ε, περισσότερο όλους για να προσανατολίζονται από το νομικό πλαίσιο. Τώρα για τις μελέτες αντικτύπου. Οι μελέτες αντικτύπου πρέπει να γίνονται όταν αλλάζει η ουσία, η βασική αρχή, όταν ε, προσθέτει ε, προτείνεται κάτι ακόμα. Όταν αντανακλώνται οι ίδιες αρχές της προηγούμενης νομοθεσίας σε ένα ενιαίο κείμενο, εδώ δεν έχουμε καμία αλλαγή ώστε να χρειάζεται να δούμε τον αντίκτυπο. Ελπίζω ότι απάντησα σε όλα σας τα σχόλια. προτείνω να γίνει μια σύγκριση με υφιστάμενα νομικά πλαίσια, τι υπήρχε, τι αλλάζει και θα δείτε ότι όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι βασικές αρχές ε, παραμένουν οι ίδιες. Ευχαριστώ. Ωραία, ωραία. Μας καθησυχάζει αυτό, δηλαδή που λέτε ότι είναι απλούστευση και εισαγωγή κανόνων ισότητα και, και από την πριν είχαμε τέσσερις οδηγίες και τώρα ένα κανονισμό. Γιατί πάντα υπάρχει ένας μικρός φόβος σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι δηλαδή μπορεί να υπάρξουν απόπειρε εισαγωγή και προσθήκη και άλλων λύσεων σε, ένα τέτοιο, σε μια τέτοια πράξη. Ε, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά προσεκτικά. Η διατήρηση των σπάνιων βόηων φυλών είναι πολύ σημαντικό εις ό,τι αφορά την παράδοση αλλά και τη γενετική. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό λοιπόν για τις περιφέρειές μας. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης που αφορά εν μέρη το προηγούμενο. Είναι οι παραπομπές στη ζωοτεχνική νομοθεσία. Εδώ η πρόταση αποσκοπεί στο να παλύψει τις αναφορές στην ζωοτεχνική νομοθεσία των οδηγιών 89 κάθετος 608, 90 κάθετος 425 και 91 κάθετος 496. Ε, αυτή η πρόταση είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και είναι η άμεση συνέπεια της πρότασης Επιτροπής ε, ε, για ένα κανονισμό σχετικά με τους επίσημους ελέγχους. Εδώ έχουμε τη γνωμοδότηση της Μπρίτα Ράιμερς. Εκείνη ήταν η συντάκτρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στην πρώτη ανάγνωση το κείμενο στις 15 Απριλίου και περιμένει τώρα την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Ζητώ τον, από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να λάβει το λόγο ή δεν χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Σαμίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν χρειάζεται ουσιαστικά να μιλήσω γιατί το κάλυψα το θέμα πριν. Είπα ότι είναι τεχνική η τροποποίηση που αφορά την προηγούμενη πρόταση και ε, πρέπει να υπάρχει ούτω ώστε να υπάρχει νομική ασφάλεια από τώρα μέχρι που θα εγκριθεί η πρόταση και μέχρι ότου ε, εγκριθεί ο καινούριος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα μεταβατικό διάστημα που θα καλύπτει τους επίσημους ελέγχους. Αυτό επιτυγχάνεται με αυτό το τεχνικό μέτρο. Ευχαριστώ πολύ. Και μετά από αυτές τις διευκρινήσεις τελειώνουμε με το σημείο αυτό. Και μπορούμε να πάμε στο ε, τελευταίο θέμα πριν από τη συνάντηση με τον Ιταλό Υπουργό. Κλωνοποίηση βοηδών, χειροειδών, προβατοειδών, εγωειδών και υποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς. Η πρόταση αυτή σκοπό έχει να αναστείλει την τεχνική και την ε, εμπορία κλώνων ζώων και εμβρίων και ο στόχος ε, που στηρίζεται στο κανονισμό 43.2 του Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διασφαλίσει ενιαίους όρους ε, και να προστατεύσει την υγεία και την καλή μεταχείριση και κατάσταση των ζώων. Επίσης η πρόταση αυτή νομιμοποιείται από τα προβλήματα για την καλή διαβίωση των ζώων που αφορούν την κλωνοποίηση και το, την αναφορά στο σημείο 13 της συνθήκης. Ε, η, στην προηγούμενη θητεία η νομοθετική πρόταση για τα νέα τρόφιμα που αφορούσαν και τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Ακόμα και στη φάση της συνδιαλλαγής, οι απόψεις ε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κλωνοποίηση παρέκλειναν υπερβολικά και έτσι δεν μπόρεσε, να καταλήξει, δεν μπόρεσε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής να καταλήξει κοινό κείμενο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες προτάσεις διαχωρίζοντας το θέμα της κλωνοποίησης από την νέα πρόταση που κάνει η Κομισιόν για τα νέα τρόφιμα. Εγώ θα συνιστούσα να έχουμε υπόψη μας αυτή αυτό το ιστορικό όταν αναλύουμε τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είναι σημαντικές πληροφορίες γιατί αντικατοπτρίζουν τη βούληση της Επιτροπής και των Ευρωβουλευτών από την προηγούμενη θητεία. Και επίσης έχουμε μια ανεπίλητη σύγκρουση αρμοδιοτήτων με την Επιτροπή Περιβάλλοντος που προσέβαλε την ανάθεση αυτού του φακέλου στην Επιτροπή μας. Πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή, προτείνω να εξετάσουμε παράλληλα και τη συναφή πρόταση εμπορίας τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα, που είναι το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας. Λοιπόν, προτείνω να συνδυάσουμε τις δύο αυτές προτάσεις. Και πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή θα ήθελα να πω ότι προτείναμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να χωρίσουμε μεταξύ μας τις δύο ονομοδοτήσεις. Η πρώτη είναι πολύ κοντά σε μας γιατί έχει να κάνει με την αναπαραγωγή. Αυτό λοιπόν θα το χειριστεί η δική μας η Επιτροπή και η δεύτερη γνωμοδότηση σχετικά με την εμπορία των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα που αφορά περισσότερο την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Αυτή η γνωμοδότηση λοιπόν να γίνει από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ακόμα δεν μας είπαν τι πιστεύουν, δεν ξέρουμε τι θα πούν, αλλά αυτό ε, είναι μια συμβαστική πρόταση. Δίνω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, προχωρήστε στη δήλωσή σας. Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που συνδυάζετε τα δύο αυτά σημεία διότι είναι αλληλένδετα. Παρά το γεγονός ότι βασίζονται σε διαφορετικά άρθρα της συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δύο οδηγίες. Η μία βάσει του άρθρου 43 της ε, συνθήκης και προτείνει την απαγόρευση χρήσης ε, τεχνικών κλωνοποίησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σκοπούς γεωργίας και ταυτόχρονα απαγορεύει και την εισαγωγή ζωντανών κλώνων για εκτροφή ε, από τρίτες χώρες. Η δεύτερη πρόταση βασίζεται στο άρθρο 352 της συνθήκης, η οποία απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά οποιονδήποτε τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Θα ήθελα να διευκρινίσω εδώ ότι αυτό το οποίο δεν καλύπτεται στις προτάσεις είναι η κλωνοποίηση για άλλους σκοπούς. Παραδείγματος χάρη έρευνα, κλωνοποίηση για ιατρικούς ε, σκοπούς, ε, για ιατρικές συσκευές ε, ή για ψυχαγωγία. Αυτό λοιπόν σχετίζεται μόνο με την ε, κλωνοποίηση για τη γεωργία και την κτηνοτροφία και συνεπώς για παραγωγή τροφίμων. Θα πρέπει να ε, πω επίσης ε, κάτι το οποίο συνάδει και με την πρόταση του Προέδρου να χωριστεί σε δύο τμήματα αυτή η νομοθεσία. Αυτό δεν βασίζεται καταρχήν για λόγους, σε λόγους ασφάλειας τροφίμων, διότι οι λόγοι για την απαγόρευση των τεχνικών κλωνοποίησης και της εισαγωγής ε, κλωνοποιημένων τροφίμων ε, έχουν σχέση με τα θέματα τα οποία αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Ασφάλειας των τροφίμων ε, και θεωρεί ότι έχουν να κάνουν με την ευημερία των ζώων. Γνωρίζουμε την ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, το Ευρωβαρόμετρο μας λέει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι αυστηρά κατά της κλωνοποίησης και επίσης ε, έχουμε υπάρξει και μάρτυρες σε προηγούμενες συζητήσεις για τα νέα τρόφιμα αυτού του γεγονότος και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να τα εξετάσουμε ξεχωριστά. Η πρόταση είναι πολύ απλή και βασίζεται σε πολύ ε, σαφώς καθορισμένους ορισμούς για το τι είναι τεχνική κλωνοποίηση και τι είναι κλωνοποιημένα τρόφιμα ή τρόφιμα τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα προϊόντα. Προτείνονται η απαγόρευση των, της εισαγωγής ζωντανών κλώνων και η απαγόρευση διάθεσης της αγοράς ε, προϊόντων τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να περάσουμε τώρα στις ε, παρεμβάσεις ε, των ε, συναδέλφων. Η κυρία Γιούσο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο διότι ήμουν σκιώδης εισηγήτρια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο κανονισμό για τα νέα τρόφιμα, τα οποία περιλάμβαναν και κρέας το οποίο προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα. Θα ήθελα να πω το εξής μπορούμε να απαγορεύσουμε ή να μην απαγορεύσουμε. Αυτό είναι ανεξάρτητο από την απόφαση των νομοθετών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να ισχυριστούμε αυτό το οποίο ε, παρουσιάστηκε ως ισχυρισμός, δηλαδή το να προσπαθήσουμε να εχνηλατήσουμε όλα τα ζώα τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ε, σε όλες τις γενναίες. Ε, αυτό είναι αδύνατο πρακτικά και δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους κτηνοτρόφους να κάνουν αυτή την ιχνηλάτηση. Καταρχάς διότι πρακτικά είναι αδύνατο, διότι είναι πάρα πολλές οι γενναίες και επίσης διότι αυτό ο οποίος ελέγχει δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό. Επομένως ε, πολύ καλά το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιτάχθηκαν σε αυτό, γι' αυτό ακριβώς και δεν έγινε αποδεκτό και δεν ε, καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στη διάρκεια της συνδιαλλαγής. Έχουμε αυτή τη στιγμή ενώπιον μας και τις ε, δύο προτάσεις και για τα νέα τρόφιμα και για τα κλωνοποιημένα ζώα και εδώ συμφωνώ απολύτως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν δεν θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε κλωνοποιημένα ζώα και να χρησιμοποιούνται τεχνικές κλωνοποίησης, θα πρέπει να το απογορεύσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να πετούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Τίποτα άλλο. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και ε, ελπίζω όλα να καταλήξουν σε αίσιο Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιούζο. Θα ήθελα να ξέρω ποιοι θέλουν το λόγο καταρχάς για να μπορέσουμε να δούμε λίγο και πόσο χρόνο ομιλίας θα έχει ο καθής. Να σας πω ότι στις 11.30 θα πρέπει να ολοκληρώσουμε με το σημείο αυτό, διότι να σας υπενθυμίσω ότι εκείνη την ώρα θα έρθει ο Υπουργός ε, Γεωργίας, ε, ε, ο Ιταλός Υπουργός Γεωργίας, Ε, η κυρία Χάουσλινγκ, δύο ή τρία λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Ο κύριος Χάουσλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η τρια λεπτα ο καθενα παρακαλω ο κυριο χαουσλινγκ λύση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να πετύχει να χωρίσουμε τις αρμοδιότητες, αλλά από την πλευρά μας πρέπει να πούμε ως άγκρι ότι η τεχνική κλωνοποίηση ε, δεν είναι καλή, όχι γιατί δεν αρέσει μόνο στους πολίτες, αλλά γιατί δείχνει προς μια ε, συγκεκριμένη κατεύθυνση της ε, ζωικής παραγωγής. Δεν τη χρειαζόμαστε αυτή την ε, ε, κατεύθυνση όχι μόνο για λόγους αρχής και ηθικής, αλλά και επειδή πιστεύουμε ότι δεν έχει νόημα να εισαχθούν τέτοιες τεχνικές. Υπάρχει ένα θέμα στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην αποτυχία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Δηλαδή, δεν πρόκειται μόνο για ζώα που κλωνοποιούνται για να μπουν στην αγορά, αλλά και τα εκτρεφόμενα ζώα, των οποίων το κρέας θα πάει στην αγορά. Τώρα αυτά θα πρέπει να αναγράφονται και στις εισαγωγές. Εδώ δημιουργείται πρόβλημα. Και θα πρέπει να το συζητήσουμε ε, ευθέως όταν ε, διαπραγματευόμεθα με τους Αμερικανούς που δεν έχουν σήμανση στο βαθμό που ε, δεν έχει ρυθμιστεί αυτό το θέμα θα υπάρχουν φόβοι ότι θα υπάρχουν κλωνοποιημένα ζώα στην ευρωπαϊκή αγορά ή αναπαραγωγικό υλικό τους χωρίς σήμανση. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι Ευρωπαίοι δεν το δέχονται αυτό. Θα πρέπει να έχουμε σαφή προστασία των Ευρωπαίων Γεωργών αλλά και του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Δηλαδή δεν θέλουμε να προωθήσουμε μέσω εισαγωγών μιας τεχνολογίας που την απορρίπτουμε στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και στο μυαλό μας και στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ γιατί υπάρχουν βασικές διαφορές ε, σε μια τεχνολογία που απορρίπτουμε. Και αυτό Νομίζω ότι δεν το έχει καταλάβει η Κομισιόν ότι δεν πρόκειται μόνο για τα κλωνοποιημένα ζώα αυτά καθ' αυτά, αλλά και για τις μεθεπόμενες γενναίες που πρέπει να σημαίνονται και να ε, αποσυρθούν από την αγορά. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να τα έχουμε. Και πρέπει να είναι σαφές ότι εμείς ε, μαζί με τους ε, παραγωγούς, τους εκτροφείς και τους πολίτες θα απορρίπτουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως ε, το γνωρίζει πλήρως αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Άντριου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την άποψή μου. Όπως είπε και προλαλή σας, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και η νομοθεσία που μας προτείνει είναι ανεπαρκής. Εάν ε, δούμε ε, λίγο τις λεπτομέρειες, θα δούμε ότι δεν ε, απαγορεύουμε σε καμία περίπτωση τα τρόφιμα τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και μπορούν τελικώς να εισαχθούν αυτά. Δεν υπάρχει καμία ετικέτα, καμία εχνηλασιμότητα του αναπαραγωγικού υλικού και δεν μπορούμε να πάμε πέραν της πρώτης γενεάς. Και επίσης δεν προβλέπεται ετικετοθεσία και για τα τρόφιμα τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Που σημαίνει ότι στην ουσία πέραν μιας γενικότερης ε, ε, απόρριψης της αρχής θα πρέπει στον κανονισμό αυτό να προσπαθήσουμε να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι διότι οι προτάσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την άποψή μου δύσκολα μπορούν να γίνουν αποδεκτές διότι περιλαμβάνουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να δεχτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ehm, er Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγα χρόνια το θέμα συζητήθηκε στα πλαίσια του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα. Τότε ήμουν στην Επιτροπή μας εγώ εισηγητής. Εκπροσώπησα την Επιτροπή μας μάλλον στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που ήταν αρμόδια επί της ουσίας. Και καθόμουν μέχρι τις 6 το πρωί στο Συμβούλιο, άσκοπα από ό,τι απεδείχθη, και έφευγα άπρακτος γιατί απετύχει ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα. Και τώρα μπαίνει το θέμα της ε, συνέχειάς της. Ε, ε, θα έπρεπε να υπάρχει κανονισμός εδώ, ούτως ώστε τα κλωνοποιημένα ζώα στην Ευρώπη ε, όχι μόνο να απορρίπτονται όπως ε, λένε οι καταναλωτές και δηλώνουν και οι γεωργοί που λένε ότι δεν τα χρειάζονται, γιατί δεν υπάρχει καμία λογική ανάγκη ε, κλωνοποίηση στη γεωργία ούτε για την παραγωγή κρέατος άλλωστε η τεχνική θα ήταν πολύ δαπανηρή και επίσης και για το αναπαραγωγικό υλικό δεν χρειάζονται το θέμα είναι οι επόμενες γενναίες εδώ ο Μάρτιν Χόισλινγκ έχει δίκιο. Βέβαια, ε, ήδη εισάγουμε από την Αμερικανική Ήπειρο και από την Νότια Αμερική και από τη Βόρεια Αμερική και από την Καναδά μεγάλες ποσότητες κρέατος και η ε, σήμανση των, ε, σχετικά με τις επόμενες γενιές θα ήταν αδύνατη. Γιατί δεν είναι το θέμα ότι είναι κλωνοποιημένη μητέρα, αλλά ο πατέρας, το α, σπέρμα δηλαδή που χρησιμοποιείται είναι από κλωνοποιημένα ζώα. Ε, αυτό επιστημονικά δεν αποδεικνύεται γιατί το σπέρμα αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με τον μη κλωνοποιημένο. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που πρέπει να μας απασχολήσει. Όλα τα άλλα ε, είχαν ε, αποφασιστεί κατά πλειοψηφία δεν έχουμε δηλαδή άλλα μείζωνα θέματα. Το μόνο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι τι θα γίνει με τους επιγενωμένους και μέχρι ποια γενεά θα κάνουμε την εξέταση και σε ποια γενιά θα πούμε ότι από εκεί και πέρα ούτε να ελέγξουμε μπορούμε, ούτε να ειχνηλατήσουμε μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λουαζό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε δίκιο οι συνάδελφοι. Όταν δεν μπορούμε να έχουμε χνηλάτιση ε, των τροφίμων, ο κανονισμός αυτός είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο στις χώρες οι οποίες ε, κάνουν κλωνοποίηση, πιο συγκεκριμένα στις Ηνωμένε Πολιτείε και εισάγονται αυτά τα προϊόντα τελικώς ε, στη εδάφη μας χωρίς να το επιτρέπει η νομοθεσία μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι πονίδιστο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τρόφιμα τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα προϊόντα. Πρόκειται για ένα κανονισμό ο οποίος επιβαρύνεται επειδή δεν θέλουμε να έχουμε ετικετοθεσία και φυσικά είναι δώρο για τους Αμερικανούς και τις μεγάλες business οι οποίοι ουσιαστικά εισάγουν προϊόντα ε, και στη Γαλλία και πραγματικά είναι σκανδαλώδες αυτό. Υπενθυμίζω ότι η κλωνοποίηση δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Ε, υπάρχει το, ε, τα πρόβλημα της ε, υγείας ε, των ζώων, υπάρχει πολύ αυξημένο κίνδυνος επιδημιών και επίσης υπάρχει και το θέμα της γενετικής διαφοροποίησης, το οποίο μπορεί να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο. Κάποια ε, είδη ε, παράγουν πολύ λίγα ζώα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μίλλερ. Κύριε Πρόεδρε, η Κομισιόν υποβάλλει εδώ μια Κομισιόν για να παρεμποδίσουμε την κλωνοποίηση στην Ευρώπη και να παρεμποδίσουμε τις εισαγωγές. Οι προλαλήσαντες συνάδελφοι έχουν καταδείξει τις αδυναμίες και σε εμά εναπόκειται να ε, ενσωματώσουμε καλύτερες προτάσεις γιατί θέλουμε βελτιωμένη προστασία των ζώων. Αυτό είναι η υψηλή προτεραιότητα στην Ευρώπη. Και ουσιαστικά η προβληματική είναι η ίδια. Είτε παίρνουμε ε, κρέας με ορμόνες και το εισάγουμε στην Ευρώπη, ε, και εκεί είναι δύσκολη η απόδειξη ή κλωνοποιημένο κρέας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε μέσα από την ε, ετικέτα, την επισήμανση να ασκήσουμε επιρροή. Και χαίρομαι διότι εδώ υπάρχει η ε, πρόθεση παρεμπόδιση στον, ειδικό κανονισμό χωρίς να ενσωματωθεί το θέμα στον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα. Ευχαριστώ πολύ. Het is echt erg zorgelijk wat hier gebeurt. We zien hier nu twee Ευχαριστώ πολύ. Είναι ανησυχητικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχουμε δύο οδηγίε, δύο οδηγίες ε, οι οποίες αφορούν διάφορα είδη και προϊόντα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για όλα τα δίδη. Παραδείγματο χάρη περιοριζόμαστε μόνο στα εγωιδή, ε, στα ε, ε, χοιρινά, στα βοηδή και αυτά σε κάποια πλαίσια. Παραδείγματο χάρη σε γεωργικό πλαίσιο. Υπάρχουν όμως άλλα προϊόντα τα οποία αποκλείονται από τις δύο οδηγίες και δεν καλύπτονται από την απαγόρευση που βλέπει είτε η μία οδηγία είτε η άλλη. Παραδείγματο χάρη τι γίνεται με τα ε, νεκρά ζώα. Ε, τα πάντα αναφέρονται σε ζώντα ζώα. Τι γίνεται επίσης ε, με τα ε, ε, μικρά ζώα τα οποία θα εισαχθούν και μετά δεν θα υπάρχει ετικετοθεσία. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν με αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε λοιπόν ε, συγκεκριμένα ζώα ε, ούτε τα, ε, τους απογόνους στη συνέχεια ε, πρέπει όλα αυτά να τα διευκρινίσουμε, διότι τα μέτρα είναι συμβολικά. Έχουμε αποκλείσει πολλές περιπτώσεις. Κατά την άποψή μου λοιπόν θα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, θα υπάρχουν προβλήματα για παράδειγμα ε, με θέματα εκτροφής και ε, θεωρώ ότι δεν είναι πραγματικά ουσιαστικό αυτή η νομοθεσία, είναι απλώς συμβολική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Όταν αυτή η οργάνωση, όπως και να αποκαλείται, είχε πει ότι όλα αυτά γίνονταν για το όφελος των ανθρώπων. Λένε το ότι οι καταναλωτές το θέλουν, δεν το χρειάζονται και οι γεωργοί. Τελικά ποιος θα υποφεληθεί από αυτό. Συνεχίζουμε να ακούμε για νέες τεχνολογίες που ε, θα θρέψουν ε, τους ανθρώπους. Θα ε, σταματήσουμε όμως τους πολεμούς, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει. Εδώ μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις, πώς μπορούν να ελέγξουν τις προμήθειες των τροφίμων, την προσφορά των τροφίμων ε, και ε, θα δημιουργήσει στην Ιρλανδία αυτό το θέμα μεγάλο ζήτημα. Ε, εγώ θεωρώ ότι ε, πρέπει να δούμε τι λέει και το ευρωβαρόμετρο, ότι δεν το θέλουμε. Μπορεί να έχουν δίκιο, μπορεί να έχουν άνθρωποι αλλά πρέπει να το πουλήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και δεν το θέλουν. Πρέπει να τους ακούσουμε αφού δεν το θέλουν, ε, να μην το κάνουμε. Είναι πολύ απλό. Αν ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ε, λαούς, ε, θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιάκοβιτς. Ευχαριστώ. Είμαι κατά της κλωνοποίησης και κατά της χρήσης κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα. Η Ευρώπη έχει ένα πολύ καλό σύστημα ελέγχου της προέλευσης των τροφίμων και της ποιότητας των τροφίμων. Έχει ένα πολύ καλό σύστημα ετικετοθεσίας. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι το ελάχιστο για το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ένα καλό σύστημα σήμανσης των κλωνοποιημένων προϊόντων. Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα χρωματικό κώδικα παραδείγματο χάρη και αυτό θα ήταν πολύ απλό έτσι ώστε να καταλαβαίνουν οι καταναλωτέ αμέσω ότι πρόκειται για κλωνοποιημένο, για κρέα από κλωνοποιημένα ζώα. Εγώ προσωπικά θα ήμουν ε, υπέρ μια τέτοια ε, επιλογής, αν είχαμε μια τέτοια ετικέτα στο, στο πακέτο του κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα, Νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε ετικέτες, να υπάρχει σήμανση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πετήλ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ε, η διάθεση μόνο από κλωνοποιημένα ζώα στην αγορά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν πρόκειται εδώ για επίλυση ενός προβλήματος επισητιστικού, αλλά πρόκειται για ένα πολιτικό θέμα. Νομίζω ότι η διάθεση τροφών από ζώα θέθεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο το δικό μας σύστημα γεωργίας και εκτενοτροφίας... Δεν φαντάζομαι ότι θα ήθελαν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να ακολουθήσουν μια τέτοια ανήθικη μέθοδο. Εγώ εκπλήσωμαι που η Κομισιόν κάνει κάποιες εξαιρέσεις καθώς εκτιμάω ότι η κλωνοποίηση δεν μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε κάποιες απτόχθονες ράτσες. Ε, χρειαζόμαστε μια τράπεζα γονιδίων. Εγώ θα πρότεινα στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής να κάνουμε μία μελέτη για να δούμε σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη ήδη έχουν δημιουργήσει τέτοιες γενετικές τράπεζες, τράπεζες γονιδίων και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο προπολογισμού για να δημιουργήσουμε τα για να διατηρήσουμε τα ήδη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριο Ντες και κατόπιν αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο έχουμε χρόνο. Παρακαλώ κύριε Ντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα και στο παρελθόν το συζητήσαμε συχνά και νομίζω ότι συμφωνήσαμε πολύ στο ότι είμαστε κατά της κλωνοποίησης. Εγώ ήμουνα 40 ε, χρόνια εκτροφέας ε, βοηδών και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει κλωνοποίηση. Τώρα έχουμε τη, δυνατότητα μεταφοράς εμβρίων που είναι άλλη διαδικασία που δεν δημιουργεί προβλήματα ηθικής. Εμείς κάναμε μεταφορά εμβρίων και η τεχνική εξαπλώθηκε γρήγορα. Δεν χρειάζονται λοιπόν οι κλόνοι γιατί δεν τους καταλαβαίνω εδώ τους Αμερικανούς. Και στην εκτροφή βοηδών υπάρχει δυνατότητα στα νεαρά ζώα να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν είναι ενδεδειγμένα για ζώα αναπαραγωγής. Δεν χρειάζεται δηλαδή να εξετάσουμε 40 ζώα για να δούμε ε, μετά από κάποια χρόνια αν ε, έχει αποδειχθεί καλό. Μετά τη γέννηση, αναλύοντας το ε, κληρονομικό υλικό, μπορούμε να είμαστε σίγουροι μέχρι και κατά 98% ότι ενδείκνεται για την εκτροφή. Οπότε η κλωνοποίηση για μένα είναι απόλυτα περιττή και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην επιτρέψουμε την εισαγωγή των ζώων αυτών εδώ σε εμά. Ένα πρόβλημα υπάρχει βέβαια αν στην Αμερική, ε, ε, στην, ε, δηλαδή αν έγινε η κλωνοποίηση πριν από 10 χρόνια, είναι δύσκολο να δούμε μετά από 10 χρόνια αν τα ζώα προέρχονται από κλωνοποίηση ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και θα πρέπει στις εμπορικές συμφωνίες μας γιατί εγώ είμαι υπέρ της σύναψης εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα πρέπει να μπουν όροι, ότι στο μέλλον οι Αμερικανοί πρέπει να έχουν σήμανση στα κλωνοποιημένα ούτω ώστε να αποκλειεται κρεας κρέα ζώων κλωνοποιημένων μετά από 5-10 χρόνια να έρθει εδώ σε εμά για το παρελθόν δεν μπορούμε να το ζητήσουμε, αλλά στα πλαίσια της εμπορικής συμφωνίας ε, εμεί πρέπει να υποβάλουμε σχετικές προτάσεις, ούτως ώστε στο μέλλον οι κανόνες να είναι καθαροί. Ευχαριστώ, κύριε Σέντρα. Κυρία. Ναι, Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με του συναδέλφου που εξέφρασαν την αντίθεσή του στην κλωνοποίηση, αλλά θέλω να αφαιρθώ σε δύο ζητήματα. Καταρχήν πιστεύω ότι η ολική απαγόρευση στην παραγωγή, θέση σε εμπορία και εισαγωγή, μηδενική ενοχή για τι επόμενε γενναίε κλωνοποιημένων ζώων, του απαγόνου δηλαδή, των κλωνοποιημένων ζώων. Και θέλω να προσθέσω ένα ακόμα επιχείρημα. Πιστεύω ότι αυτέ οι τεχνικέ οδηγούν ε, σε εξάρτηση των γεωργών ε, και είναι ένα ακόμα βήμα για την καταστροφή των μικροπεσίων γεωργών. νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την βιώσιμη γεωργία η οποία θα σέβεται και την ευημερία των ζώων. Σας ευχαριστώ. παρακαλώ. Κύριε Εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει να βάλει τα δυνατά της για να προστατεύσει την ποιότητα και την βιοπικιλότητα. Και δεν θα πρέπει να κάνει δώρα στην ήδη εντατική παραγωγή κλοπένων ζών στην Κίνα και στις Ηνωμένε Πολιτείες και το μόνο που θα γίνει είναι να οδηγηθεί σε ύφεση η ευρωπαϊκή οικονομία. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Να δώσω κατόπιν το λόγο στους εκπροσώπους της ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ. Κύριε Μίκο, παρακαλώ. Θα σας ζητούσα να απαντήσετε στις παρεμβάσεις που ακούστηκαν και αν θέλετε μπορείτε να μας δώσετε και πρόσθετες πληροφορίες. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, όπως αναμενόταν. Το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ σημαντικό. Και είχα το προνόμιο να συμμετάσχω και στην προηγούμενη θητεία στον τριμερή διάλογο και παρακολούθησα παρόμοιες συζητήσεις και τότε. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω κάποια σημεία και να προσθέσω και κάποιες λεπτομέρειες. Αρχίζω ε, από κάτι που αναφέρθηκε ήδη από αρκετά μέλη. Η κλωνοποίηση δεν είναι γενετική τροποποίηση. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να ανοιχνευθεί με εξέταση του ατόμου. Δηλαδή δεν μπορεί να βρεθεί αν το άτομο κλωνοποιήθηκε ή όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι δεν έχουμε στα χέρια μας αντικειμενική μέθοδο ελέγχου. Ο μόνος τρόπος ελέγχου είναι επιχάρτου δηλαδή με την ιχνηλασιμότητα με βάση ε, τις καταχωρήσεις που έγιναν και την Τράπεζα Ιχνηλασιμότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την επισήμανση των ίδιων των κλώνων ή των ε, απογόνων της τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενεάς. Στην πράξη είναι αδύνατον να το ελέγξουμε αυτό στις επόμενες γενιές. Και αν επιμένετε να δημιουργηθεί σύστημα που θα παρακολουθεί τις επόμενες γενιές, θα φτιάξετε ε, ε, ένα, ε, ένα μηχανισμό δαπανηρό και σούπερ γραφειοκρατικό. Εμείς κάναμε κάποιες αξιολογήσεις και καταλήξαμε ότι το κόστος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μιλάω μόνο για το κόστος των Αμερικανών εκτροφέων που χρησιμοποιούν κλόνους, όπως ε, θεωρήσατε στη συζήτηση αυτή. Αυτό είναι κόστος για τους Ευρωπαίους ε, ε, εκτροφείς που πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν κλόνους με το ίδιο σύστημα. Δηλαδή όλη αυτή την ευρεία καταχώρηση και θα πληρώνουν το κόστος ε, για τα βοηδή τους τρίτης τέταρτης γενιάς. Εμείς έχουμε ένα καλό σύστημα επισήμανσης, ιδιαίτερα για τα βοηδή στην Ευρώπη, όχι τόσο για τα άλλα. Αλλά εδώ πρόκειται για πρόσθετες προσπάθειες, πρόσθετο κόστος και επαναλαμβάνω. Τυπικά είναι πιθανό, είναι δυνατόν, αλλά στην πράξη δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Γιατί το γενετικό περιεχόμενο του ατόμου είναι ακριβώς το ίδιο όπως το πρωτότυπο και δεν θα ανοιχνεύσετε αλλοιώσεις, αλλαγές ή τροποποίησεις. Παρ' όλα αυτά όμως το σκεφτόμαστε και ε, πρέπει να το πω αυτό ξεκάθαρα γιατί άκουσα στη συζήτηση ότι θα έρθουν οι εισαγωγέ κλώνων από τις ΙΠΑ, θα τρώμε τα κλωνοποιημένα κρέατα. Όχι. Ακριβώς αυτό είναι που απαγορεύεται από την πρόταση. Απαγορεύομαι τις εισαγωγές των κλώνων και απαγορεύομαι η αδίποτε τρόφιμα από τους κλώνους. Μικρή τεχνική λεπτομέρεια. Κάντε μια διάκριση παρακαλώ. Δεν υπάρχει κλωνοποιημένα τρόφιμα, δεν υπάρχουν κλωνοποιημένα, τα τρόφιμα δεν κλωνοποιούνται, το ζώο κλωνοποιείται και μετά θα φάτε τα τρόφιμα από το κλωνοποιημένο ζώο. Δεν υπάρχουν όμως κλωνοποιημένα τρόφιμα. Αυτό τεχνικά είναι αδύνατον. Όταν συζητήσαμε την τελευταία φορά το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, το θέμα ήταν η επισήμανση των απογόνων των υπομένων γενεών, αλλά το αποτέλεσμα της συζήτησης ε, ήταν ότι αναφέρθηκαν τα κόστη και η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν θεώρησε ότι ήταν τόσο μεγάλα και αποφάσισαν να αξιολογηθεί η πρόταση λεπτομερώς πριν δοθεί συνέχεια. Η δική μας αξιολόγηση και εκτίμηση που κάναμε πριν υποβάλουμε την πρόταση δείχνει ότι το κόστος είναι υπερβολικό. Αλλά οι επίτροποι αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερο και για τις δικές σας συζητήσεις ε, θα ήταν καλύτερο να υπάρχει μία σε βάθος ανάλυση. Η ανάλυση συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες. Οπότε θα έχουμε και συμπληρωματικά στοιχεία για το, τα συναφή κόστη, συναφή με τη, τους κλόνους. Να πω ακόμη ότι όταν μιλάμε για τις δυνα... πιθανές εξαιρέσεις, ε, πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει εξαίρεση για κλόνους ε, που αφορούν την παραγωγή τροφίμων ή την ζωική παραγωγή. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι μοναδικές εξαιρέσεις αφορούν την ιατρική, την επιστήμη, την ιατρική και την ε, διατήρηση των κονοτύπων που μας επιτρέπει να διατηρήσουμε το τελευταίο ζώο αυτού του γονότυπου αν δεν έχουμε άλλο μέσον. Δεν ε, θα ήταν καλή κίνηση να μην επιτρέψουμε την, τις περαιτέρω εξελίξεις αυτούς τους τομείς και διότι ε, θέλουμε ε, να προωθήσουμε την ιατρική και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα εδώ παίζει ρόλο η κλωνοποίηση και η κλώνη Γι' αυτό περιοριζόμαστε στους κλόνους στην ζωική παραγωγή, στις εκμεταλλεύσεις και στα τρόφιμα. Αναφέρθηκε επίσης ότι μπορεί να δημιουργηθεί εξάρτηση των ε, εκτροφέων και άκουσα και μια, ε, ένα παραλληλισμό με τους σπόρους. Τα δύο θέματα είναι τελείως διαφορετικά. Ακόμα και αν κάποιος ε, ταχθεί υπέρ της κλωνοποίησης, αναφέρθηκα και αυτό από τα μέλη, η κλωνοποίηση σήμερα και για πολύ καιρό στο μέλλον θα συνεχίσει να είναι πολύ δαπανήρη διαδικασία. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Και σίγουρα δεν δημιουργεί η αδίποτε εξάρτηση ε, των άλλων κρίκων της αλυσίδας. Αν εμείς δεν επιτρέψουμε εισαγωγή κλώνων και αν δεν επιτρέψουμε τεχνικές κλωνοποίησεις, κανένας εκτροφέας δεν θα ε, αποκτήσει εξάρτηση ε, κατιονδήποτε τρόπο από την τεχνική κλωνοποίηση. Δεν υπάρχει πίεση να χρησιμοποιούνται κλόνοι. Μπορεί να γίνεται μια συζήτηση αν κάποιος θέλει να το κάνει. Εμείς όμως λέμε σαφές όχι, ένα σαφές όχι στην Ευρώπη. Αυτά τα λέω για να απαντήσω στα περισσότερα σχόλιά σας. Θα συνεχιστεί η συζήτηση, θα είναι και περίπλοκη, σύνθετη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα πούμε αυτά τα βασικά γιατί μιλάμε για πολλές δαπάνες, μεγάλο γραφειοκρατικό μηχανισμό και για τους Ευρωπαίους ε, και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οπότε αυτό να το λάβετε υπόψη σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες και για τις απαντήσεις που δώσατε στα μέλη. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση ε, επί του σημείου αυτού σήμερα. Προφανώς θα επανέλθουμε αργότερα ε, σε άλλες περιστάσεις και στην Επιτροπή μας και στις συζητήσεις με τους ψηφοφόρους μας. Όπως σας είπα, ε, η συζήτηση για σήμερα ολοκληρώθηκε και μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα πεντάλεπτο επειδή ε, περιμένουμε να έρθει ο Ιταλός Υπουργός ε, της Γεωργίας που εκπροσωπεί την Προεδρία. Παραμείνατε στην αίθουσα παρακαλώ για να τον με όταν έρθει και να, το, να ακούσουμε τη σημαντική ομιλία του. Πέντε λεπτά διάλειμμα λοιπόν και ελπίζω να μπορέσουμε να αρχίσουμε έγκαιρα ή και πριν από το πεντάλεπτο.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 coordinators Παρακαλώ, μην με αναγκάζετε να χτυπώ τόσε πολλέ φορέ το σφυράκι μου, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ στην Επιτροπή μας Να καλωσορίσουμε λοιπόν εδώ στη συνεδρίαση τον κύριο Μαουρίτσιο Μαρτίνα, Υπουργό Γεωργίας ε, της ε, Ιταλίας, ε, που αυτή τη στιγμή έχει τα ενία της Προεδρίας του Συμβουλίου, ο οποίος είναι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου Γεωργίας. Θα ήθελα λοιπόν να μας παρουσιάσει τώρα τις ε, προτάσεις. για τα θέματα γεωργίας. Φαντάζομαι ότι θα αναφερθείτε και στις συγκεκριμένε προτάσεις της Ιταλικής Προεδρίας ε, σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη στιγμή δεδομένου ότι θα έχουμε και την ε, επιλογή των νέων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ ε, για την επιλογή της είπα εκπροσώπου η οποία είναι ε, σύντροφος του Υπουργού, η νέα ύπατη εκπρόσωπος και επίσης να πω ότι Ε, οι διάφορες ε, συζητήσεις που γίνονται σε εμπορικό επίπεδο για την αλλαγή των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα ευρωπαϊκά ζητήματα τα οποία είναι όλο ένα και πιο σημαντικά. Ε, γνωρίζουμε ότι είναι όλο ένα και πιο παγκόσμια τα θέματα τα οποία απασχολούν την Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, ε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για αυτή την σημαντική ευκαιρία που μου επιτρέπει να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασίας της Ιταλικής Προεδρίας. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω διότι με τη συγκεκριμένη συνάντηση μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα πρώτο σημαντικό διάλογο για τα θέματα τα οποία θα μας ε, απασχολήσουν ε, από τις επόμενες ημέρες. Το έργο της Επιτροπής σας είναι ζωτική σημασίας για το Συμβούλιο και σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε ευθύ εξ αρχή ε, μια πολύ έντονη και επικοδομητική αντιπαράθεση για όλα τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Από πείρα γνωρίζουμε ότι όταν τα τρία θεσμικά όργανα της Ένωσης ε, εργάζονται αποτελεσματικά και αρμονικά, τα αποτελέσματα είναι στο ύψος των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή η απόδειξη η πρόσφατη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής η οποία ε, προέκυψε στην ε, προηγούμενη θητεία με έντονες και ποιοτικά ε, εργασίες μέσω της συνεργασίας των τριών θεσμικών οργάνων και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Πάολο Ντεκάστρο για το εξαιρετικό έργο του και σε αυτό αλλά και σε άλλα ζητήματα. Θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω τα ουσιαστικά ζητήματα του προγράμματος εργασίας της Ιταλικής Προεδρίας για τον τομέα της γεωργίας, ε, πρόγραμμα στο οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες μας από τον Ιούλιο. Θα ήθελα Καταρχήν, να ε, υπογραμμίσω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργική πολιτικής ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία για το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πλέον πρέπει να συνεχίσουμε για να καθορίσουμε ε, τις ε, βασικές πράξεις που θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε την όλη διαδικασία της μεταρρύθμισης. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στις πράξεις κατεξουσιοδότηση που προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σκοπεύουμε να ολοκληρήσουμε την εξέταση αυτών των πράξεων στις επόμενες εβδομάδες. Από πλευρά Συμβουλίου δεν διαπιστώνουμε ιδιαίτερες δυσκολίες και ελπίζουμε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε ε, γρήγορα αυτές τις ε, πράξεις. Ε, μεταξύ των θεμάτων τα οποία εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα οποία θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση και μαζί σας, θα πρέπει σίγουρα να αναφέρουμε και την πρόθεση του κανονισμού για τη μεταρρύθμιση της βιολογικής γεωργίας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα ευαίσθητο για όλα τα κράτη-μέλη η βιολογική γεωργία είναι ένα τμήμα ε, αυξανόμενης σημασίας ε, ε, σε στρατηγικό επίπεδο για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας και σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια έντονη και επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι το καλύτερο δυνατό από όλες τις πλευρές και όπως γνωρίζετε μετά από την παρουσίαση της πρότασης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τεχνικό επίπεδο το Συμβούλιο έχει ήδη κάνει μια εξέταση ε, των δύο τρίτων περίπου του κανονισμού. Εν τω μεταξύ το Συμβούλιο ε, του, Ιουλίου, το πρώτο στο οποίο προείδρευσα, οι Υπουργοί μπόρεσαν να εκφράσουν και την προκατακτική τους άποψη στα πλαίσια μιας πολιτικής συζήτησης για τα βασικά ζητήματα του κειμένου. Πρόκειται για μια διαδικασία αναθεώρησης της νομοθεσίας. Ε, στα πλαίσια ε, των συναντήσεων υπήρξαν και κάποιες επικρίσεις για κάποιες πτυχές της πρότασης βεβαίως. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τη συνεργασία σας προκειμένου να ε, προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ απόψεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερο το θέμα αυτό. Εάν ε, η πορεία των διαπραγματεύσεων μας το επιτρέψει θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε να συζητούμε ένα συμβαστικό κείμενο της Προεδρίας. Ένα άλλο κείμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο αφορά την αναθεώρηση του καθεστώτος των ενισχύσεων για την ε, ε, κατανομή των ε, φρούτων και, και του γάλακτος ε, στα σχολεία. Εδώ θα συνεχίσουμε τα όσα έχει ήδη κάνει η Ελληνική Προεδρία, ωστόσο όπως ήδη γνωρίζετε όλο το Συμβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερες επιφυλάξεις για την νομική βάση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να προοδεύουμε στην πρόταση αυτή και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε ήδη καθορίσει μία σειρά από πολύ σημαντικέ συνεδριάσεις ομάδων εργασίας στο Συμβούλιο στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής Γεωργίας. Θεωρούμε ότι ε, θα πρέπει για το θέμα αυτό να γίνουν οι μέγιστε δυνατέ προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες την καλύτερη λειτουργία ενός συστήματος το οποίο θα πρέπει να συνδυάζει ταυτόχρονα την ε, ε, ε, προσέγγιση των πολιτών με το γεωργικό κόσμο αλλά και τις κατάλληλες πτυχές βελτίωσης της υγείας. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει και για το θέμα αυτό να ξεκινήσουμε συζητήσεις μαζί σας στους επόμενους μήνες με αποτελεσματικό και οργανικό τρόπο. Στόχος μας είναι να έχουμε μια γενική προσέγγιση η οποία θα μπορέσει να μας βοηθήσει στο μέλλον να επιταχύνουμε τους χρόνους και να μπορέσουμε να έχουμε ένα συμβιβασμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων ώστε να έχουμε έγκριση του κειμένου. Ένα άλλο θέμα σημαντικό είναι το θέμα του μέλλοντος του γαλακτοκαμικού τομέα. Στο θέμα αυτό, όπως είναι γνωστό, η συζήτηση σε όλα τα επίπεδα είναι μεταξύ των θεσμικών οργάνων ε, και έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την έκθεσή της για την κατάσταση του κλάδου και ε, τη δέσμη μέτρων για το γάλα. Το Συμβούλιο έκανε μία συζήτηση όπου συζητήθηκε η έκθεση αυτή και ε, γνωρίζουμε πόσο σημαντικά και ευαίσθητο είναι το θέμα αυτό, όπως επίσης θεωρούμε ότι ο γαλακτοκομικός τομέας είναι ένας στρατηγικός τομέας, θεμελιώδης ε, τομέας πρώτης γραμμής. Η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και το γαλακτοκομικό πακέτο μας ε, έδωσαν τη δυνατότητα να έχουμε κάποια νέα στοιχεία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση της αγοράς και να βελτιώσουμε τη λειτουργία όλης της αλυσίδας διανομής. Ωστόσο, η Προεδρία γνωρίζει ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το θέμα αυτό, ε, διότι από του χρόνου θα πάυσει το καθεστώς των ε, ποσοστώσεων και επομένως θα παρακολουθούμε ιδιαίτερα προσεκτικά την κατάσταση. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας, αφορά την ε, επισητιστική ασφάλεια, το πιο περίπλοκο ζήτημα και σε θέμα ε, κατάλληλης διάθεσης τροφίμων αλλά και της ισότιμης ε, διανομής του. Καθώς επίσης και να υπάρχουν και στρατηγικά ε, εφόδια γεωργικών πρώτων υλών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο συζητούμε εδώ και αρκετό καιρό σε όλα τα επίπεδα, σε όλο τον κόσμο και πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις στο μέλλον ε, και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο κλειδί στην πρώτη γραμμή. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες και θα προσέξουμε ιδιαίτερα. Το θέμα θα βρίσκεται και στο επίτροπο της Παγκόσμιας Έκθεσης του Μιλάνο ε, το 2015 που έχει ένα εξαιρετικό τίτλο ε, θρέφουμε τον πλανήτη, ενέργεια για τη ζωή. Και πέραν ε, της εξαιρετικής αυτής εκδήλωσης ε, για όλο τον γεωργικό διατροφικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι και μια εξαιρετική πλατφόρμα αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, ιδιαίτερα για ένα τόσο στρατηγικό ζήτημα και για τις παρούσες προκλήσεις ε, και για τις μελλοντικές προκλήσεις, οι οποίες ε, είναι προκλήσεις οι οποίες αφορούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια σημεία κομβικά. Η Ιταλική Προεδρία σκοπεύει να θέσει το θέμα αυτό στο επίκεντρο της ε, πολιτικής συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να επικεντρώσουμε ε, την προσοχή μας στην επισητιστική ασφάλεια στη συζήτηση που θα γίνει στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας ε, στο Μιλάνο στα τέλη Σεπτεμβρίου στα πλαίσια των παγκόσμιων αυτών θεμάτων που μας απασχολούν θα πρέπει να εγγράψουμε φυσικά και τα όλα σχετίζονται με όσα σχετίζονται με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις εν εξελίξη, στις οποίες η Γεωργία έχει πολύ σημαντικό ε, ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις των διεθνών συμφωνιών και σε πολυμερές επίπεδο, ε, σε επίπεδο ΠΟΕ και στο θεματολόγιο μετά τον Παλί, αλλά και ε, σε διμερές επίπεδο θα γίνει επικαιροποίηση και συζήτηση στα πλαίσια του Συμβουλίου για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ελευθέρων συναλλαγών, ε, οι οποίες είναι εν εξελίξη, έχουν ήδη ολοκληρωθεί, πιο συγκεκριμένα τις συμφωνίες με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με τον Καναδά, τις χώρες της Ασίας, τις χώρες της Αμερικής και της Λατινικής Αμερικής και θα ε, θέσουμε στο επίκεντρο της συζήτησης τις συνέπειες και την επιρροή που μπορούν να έχουν αυτές οι ε, συμφωνίες για τον ευρωπαϊκό γεωργικό κλάδο, καθώς επίσης και την ανάγκη να υπάρχει ένα σύστημα αμοιβαιότητες επί τη βάση των συμφωνιών που θα, ολοκληρώ, ε, θα περιλαμβάνει και την αναγνώριση του ευρωπαϊκού συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων. Σε αυτό ακριβώ το πλαίσιο σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε και με την Επιτροπή σα ένα διάλογο επικοδομητικό και αντιπαράθεση. Υπάρχουν άλλα δύο θέματα τα οποία αφορούν ένα στρατηγικό όραμα για το μέλλον του γεωργικού τομέα και στα οποία η Ιταλική Προεδρία σκοπεύει να δώσει προτεραιότητα. Είναι το θέμα της αναθεώρησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της στρατηγικής για το κλίμα και την ενέργεια του 2030. Όσον αφορά την πρώτη, Σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε στον γεωργικό τομέα μία ε, εξέταση της αναθεώρησης ε, σε μεσοπρόσωπο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαρτίου. Θέλουμε να έχουμε ένα κοινό όραμα και να σκεφτούμε τις μελλοντικέ στρατηγικές μας. Πιο συγκεκριμένα η Προεδρία θα επικεντρώσει τη συζήτηση στην καινοτομία και στις ε, προοπτικές απασχόλησης των νέων γεωργών στα πλαίσια φυσικά και του Συμβουλίου Γεωργίας του Οκτωβρίου. Θα ε, υπάρξει μια συγκεκριμένη ε, συζήτηση για το θέμα αυτό. Η, το αποτέλεσμα της συζήτησης ε, θα αποτελέσει και τροφή για τις συζητήσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την αναθεώρηση της στρατηγικής και θα είναι και η συνεισφορά της Γεωργίας στη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο το Μάρτιο του 2015. Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική για το κλίμα και την ενέργεια του 2030, Αναγνωρίζουμε πλήρω τη σημασία τη μείωση ε, των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου για τον τομέα τη γεωργία, καθώ επίση και τη συνεισφορά που μπορεί να ε, προσφέρει ο γεωργικό κλάδο για να μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική μείωση. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο Γεωργίας θα κάνει μια συζήτηση επί του θέματο εν ώψη και της ε, συνεδρίασης του Οκτωβρίου και το αποτέλεσμα τη συζήτηση και σε αυτή την περίπτωση θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Περιβάλλοντο και ενέργεια τα οποία είναι τα καθήλυνα αρμόδια εν ώψη της προετοιμασίας της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα τέλη Οκτωβρίου. Είμαστε εν αναμονή τη συζήτηση λοιπόν με όλες τις αρμόδιε επιτροπέ του Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην επίτευξη αυτών των στόχων. Επίσης υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα τα οποία θα συζητηθούν στα πλαίσια της Ιταλική Προεδρίας ε, του Συμβουλίου. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση κανονισμού για τα μέτρα προστασίας για τους επιβλαβείς οργανισμούς ε, για τα φυτά, καθώς επίσης και τη δέσμη μέτρων για την νομοθεσία για, την, ε, ε, για τα ζωοτεχνικά ζητήματα. Πρόκειται για σημαντικά θέματα στρατηγικής σημασίας, τα οποία έχουν στόχο να απλωστεύσουν και το νομικό πλαίσιο, να μειώσουν το περιττό γραφειοκρατικό άκθος και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μα. Ξεκινώντα λοιπόν από αυτού του στόχου, η Ιταλική Προεδρία θα εξετάσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι προτάσει και τι τροπολογίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε επικοδομητικές ε, και καρποφόρες ε, διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για τα μέτρα προστασίας εναντίον των επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και τη δέσμη μέτρων για την ε, ζωοτεχνική νομοθεσία, αυτά θέλουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση των κινδύνων στον κλάδο λόγω της ε, εξάπλωσης ε, νέων επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών που προέρχονται κυρίως από την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και την αλλαγή του κλίματος. Ακριβώς για αυτό το σκοπό η πρόταση περιλαμβάνει νέα μέσα αξιολόγησης του φωτιογειονομικού κινδύνου καθώς επίσης και μια καλύτερη εποπτεία στις ε, επικράτειες καθώς επίσης και σε νέες αιστείες επιβλαβών οργανισμών. Ε, στο επίπεδο του Συμβουλίου κάνουμε μια τεχνική εξέταση της πρότασης βάσει της πρώτης πρότασης συμβαστικού κειμένου που ετοίμασε η Ελληνική Προεδρία. Όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για την ζωοτεχνική νομοθεσία, με τη νέα πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σκοπεύουμε να ε, έχουμε την οριζόντια ε, διάρθρωση της νομοθεσίας και όχι πλέον την κάθετη αναείδος. Θέλουμε επίσης να έχουμε συγκεκριμένες ευαίσθητες αλλαγές σε οργανωτικό πλαίσιο που φαίνεται ότι θα μπορέσουν να μειώσουν τα περιθώρια δημόσιας ρύθμισης, τα οποία φυσικά είναι πολύ σημαντικά για τα μικρά είδη τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Η Προεδρία σκοπεύει να ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση του κειμένου το οποίο προτείνεται, στα, ε, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε και το σχετικό ζήτημα και να βρούμε ποια είναι τα κοινά μας σημεία. Όσον αφορά το ευαίσθητο ζήτημα τη καλλιέργειας μη γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, τον Ιούνιο, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο Περιβάλλοντο κατέληξε σε μια πολιτική συμφωνία για την πρόταση τροποποίηση τη οδηγία για την ε, ε, εσκεμμένη εκπομπή στον, στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και η πρόταση θέλει να περιορίσει ή να απαγορεύσει οριστικά στα κράτη-μέλη ε, την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών τα οποία έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά ε, θα βασίζονται σε διαφορετικά αίτια από αυτά τα οποία προβλέπονται από, την, ε, ε, από το σύστημα το οποίο ισχύει ήδη. Η συμφωνία θα αποτελεί μια πολύ σημαντική ισορροπία μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και επομένως βάσει και της αρχής της επικουρικότητας είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα ξεκινήσουμε ως Προεδρία στις επόμενες εβδομάδες μαζί με τους συναδέλφους ε, Υπουργούς Περιβάλλοντος και Υπουργούς Υγείας θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτους. Τέλος, Επιτρέψτε μου να σταθώ σε ένα ε, πρόβλημα το οποίο ε, μας απασχολεί τις τελευταίες εβδομάδες και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αναφέρομαι στην κρίση ε, των εποχικών φρούτων και στο εμπάργο της Ρωσίας σε κάποια γεωργικά προϊόντα. Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά θέματα στα οποία η Ιταλική Προεδρία εργάστηκε ευθύ εξ αρχής, ε, ιδιαίτερα ε, εντατικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όπω είναι γνωστό ενέκρινε στα πλαίσια των εξουσιών τη ε, κάποια μέτρα για να υποστηρίξει του τομεί που χτυπήθηκαν κυρίω από αυτή την κρίση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Τσιόλο και το προσωπικό του για αυτή την αντίδραση και για τα όσα πρότεινε φυσικά. Θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω το ζήτημα και η μεταρρύθμιση τη Κυνηγή πολιτικής σε αυτό το πλαίσιο έδειξε ότι διαθέτει τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να αντιμετωπίσει κρίσεις αυτού του μεγέθους, αλλά ίσως θα έπρεπε να γίνει και μία εξέταση της ανάγκης να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτά τα μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο η ε, συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι κατά την άποψή μου ζωτική σημασία. Το έκτακτο συμβούλιο το οποίο συγκαλέσαμε για την επόμενη Παρασκευή θα μας επιτρέψει να δούμε ε, και τα μέτρα τα οποία ήδη εκρίναμε για να δούμε καθα... πόσον ε, αντιμετώπισαν την κρίση. Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι προσπάθησα συνοπτικά να σας παρουσιάσω τα βασικά ζητήματα και τα βασικά θέματα τα οποία θα συζητηθούν στα πλαίσια της Ιταλικής Προεδρίας. Είμαι φυσικά στη διάθεσή σας ε, με τους συνεργάτες μου για όλες τις πληροφορίες και τις διευκρινήσεις που ίσως θα χρειαστούν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, ε, πραγματικά ελπίζω ότι μέσω αυτής της ε, συνεργασίας θα μπορέσει να ξεκινήσει μια ε, εντατική προσπάθεια για να ξεκινήσουμε αυτό τον απαραίτητο διάλογο, ο οποίος θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτό τον τόσο ε, σημαντικό τομέα, κυρίως αυτή την ευαίσθητη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, για να μπορέσουμε να ε, κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε κληθεί να κάνουμε. Ελπίζω αυτό το επικοδομητικό πνεύμα να μας βοηθήσει στις επόμενες ώρες και εβδομάδες κοινή εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για αυτή την όσο εκτενή παρουσίαση των εργασιών της Προεδρίας. Κυρίες και κύριοι, θα να σας πω το εξή. Θα προχωρήσουμε ως εξή. Θα ακούσουμε καταρχήν τους συντονιστές, δύο λεπτά για τον καθένα. Κατόπιν θα πάρει το λόγο ο υπουργό. Ε, δεν θα ήθελα να του περιοριστώ χρόνο και κατόπιν έχουμε 20 περίπου άτομα που θα ήθελα το λόγο. Ένα λεπτό για τον καθένα για να έχουμε και τις τελικές παρατηρήσεις του κύριου Υπουργού. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην θυμώσετε όταν θα χτυπάω το σφυράκι για να μείνετε εντό του χρόνου. Το λέω γιατί στο παρελθόν κάποιος είχε θυμώσει. Στο μέλλον θα προβλέπουμε περισσότερο χρόνο για τέτοιου είδου ε, συνεδριάσεις και συζητήσεις με τους προκεκλημένους μας. Ποτέ δεν μας φτάνει ο χρόνος γιατί πάντα έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές. Ε, καταρχήν ο κύριος Ντές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ Μαρτίνα που ήρθατε στην Επιτροπή Γεωργίας. Εύχομαι και προσβλέπω σε επιτυχή συνεργασία επί της Προεδρίας σας. Ε, στα δύο λεπτά θα αναφέρω κάποια θέματα και οι συνάδελφοι άλλα. Ευχαριστώ που μιλήσατε για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις εδώ, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται στα παιδιά στα σχολεία να προσφέρουμε αυτά τα προϊόντα. ό,τι αφορά το μέλλον του, του τομέα του γάλατος, το συζητήσαμε πολύ καιρό, ε, λίγοι, λίγουν οι ποσοστώσεις ε, του χρόνου, έχουμε μια ιδιαιτερότητα εμείς και η συνάδελφος Άντρα Κορνίντε θα παρουσιάσει την κατάσταση στη Λετωνία που είναι μικρή χώρα αλλά ε, είχε πολλές εξαγωγές στη Ρωσία και θα ήθελα να μας υποστηρίξετε για την εξέβρεση λύσεων. Είναι πολύ καλό το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας που αναφέρατε και ότι χρησιμοποιήσατε στρατηγικά από θέματα. Παλιά απαγορευόταν να τα συζητούμε αυτά. Τώρα όμως πρέπει εν ώψη της διεθνούς κατάστασης να θέσουμε στο προσκήνιο το θέμα αυτό. Για τη συμφωνία με Καναδά, είπα και Νότια Κορέα, Μερκοσούρ επίσης, εδώ θα ήθελα να σας πω ότι ήδη τον Οκτώβριο του 2010 το 2000, το, στο Στρασβούργο ε, λάβαμε μια απόφαση όπου καλούσαμε την Κομισιόν να επιτρέπει εισαγωγές γεωργικών προϊόντων αν καλύπτονταν θέματα προστασίας καταναλωτών, περιβάλλοντος κλπ. Και 435 ψήφισαν υπέρ. Ε, και από την άποψη της Γερμανίας τα δικαιώματα των φυτών. Ε, θα ήθελα να μου πείτε και εδώ πώς έχει το θέμα στα δικαιώματα για τα φυτά και το αναπαραγωγικό υλικό του σπόρους. Ε, πώς θα δοθεί συνέχεια στο Συμβούλιο σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ντεκάστρο, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, αυτά τα δύο λεπτά, σε αυτά τα δύο λεπτά θέλω να υπογραμμίσω κάποια σημεία και ίσως ε, οι συνάδελφοι θα αναφερθούν σε κάποια άλλα σημεία. Κυρίως θα αναφερθώ στη διοργανική συνεργασία. Όπως ε, μας υπενθυμίσατε, είναι ένα από τα ισχυρά σημεία η μεταρρύθμιση της της ΚΑΠ ήταν ε, ένα από τα πρώτα δείγματα, από πρώτης δοκιμασίας για τη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου αλλά είδαμε και την κρίση που ξέσπασε με, την, με το ρωσικό εμπάργκο, με τη ρωσική απαγόρευση. Τώρα βλέπουμε ότι αν τα τρία όργανα συνεργαστούν σίγουρα θα έχουμε όφελος, ε, δημιουργίας ε, μία ομάδα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι έτσι αυτό θα βοηθήσει τους γεωργούς μας. Τώρα θέλω να υπογραμμίσω, Πρόεδρε, κάτι πολύ λεπτό που είναι η κατεξουσιοδότηση πράξης. Ε, εμείς θα συζητήσουμε σήμερα ε, το θέμα των ε, δικαιωμάτων φύτευσης ε, στον αμπελοϊνικό τομέα και κλεισμένων των θυρών και σε ό,τι αφορά αυτά τα δικαιώματα φύτευσης, η κατεξουσιοδότηση πράξης σημαίνουν ότι αποκλείεται το κοινοβούλιο. Εμείς μπορούμε να τις ε, απορρίψουμε. Όμως, εδώ βασιζόμαστε σε εσά γιατί για την συμφωνία συμφωνία για του, του ίνου θέλουμε να διατηρηθεί το status quo για τις χώρες που το ζητούν και δεν θέλουμε να υπάρχουν αλλοιώσεις. Τώρα σε ό,τι αφορά τη διανομή φρούτων και γάλακτος στα σχολεία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συζητήσω στο Συμβουλίο και να μιλήσουμε για ένα μεγάλο σχέδιο διατροφικής εκπαίδευσης γιατί αν εμείς απλώς μιλάμε για ένα σύστημα ε, όπου τα μόνα προϊόντα που θα διανέμονται είναι το γάλα και τα φρούτα δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτή η εκστρατεία πρέπει να είναι εκστρατεία διατροφικής εκπαίδευσης και ίσως να περιλαμβάνει και άλλα προϊόντα επίσης νομίζω ότι θα ήταν καλό να λάβει θέση η Ιταλική Προεδρία για την Εμπορική Συμφωνία με τη ΣΥΠΑ ήδη βλέπετε πόσο όλο ένα και περισσότερο να δίνονται κάποιες επικρίσεις, κάποιες ανησυχίες που είναι νόμιμες ε, φυσικά. Γιατί τα πρότυπα τετροφικά στα οποία έχουμε φτάσει εμείς θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Όμως... Όπως είπε και ο κύριος Ντες, αυτή η συμφωνία είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να εμπλακούμε στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Πρόεδρος, ο κύριος Βουτσακόφσκι, αντικαθιστά τον του κύριο Έγκερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω τρία ζητήματα. Καταρχήν ε, για το ρωσικό εμπάργο και την κρίση που πλήττει πολλές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνέπεια αυτού. Παρατηρήσαμε ότι αυτή η κρίση δεν επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό για την κρίση έτσι όπως ε, ρυθμίζεται προβλέπεται στο άρθρο 25 όπου έχουμε 400 εκατομμύρια ευρώ. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη πιο επίγουσα κατάσταση από αυτή για να χρησιμοποιηθεί αυτό το παθηματικό, κυρίως όταν μιλάμε για μια κρίση την οποία βιώνουν οι γεωργοί αυτή τη στιγμή και νομίζουμε ότι θα έπρεπε να επιβληθεί χρησιμοποιώντας τα αποθέματα αυτού του ταμείου, αυτό το παθηματικό. Θα ήθελα να εργαστεί η Ιταλική Προεδρία προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, η ε, για όσους έχουν υπερβεί τις ποσοστώσεις στον τομέα του γάλακτος. Υποτίθεται ότι αυτό ε, ήταν ε, ένα έγκλημα και τώρα κατά κάποιο τρόπο, το λέω μεταφορικά, επιβάλλονται κυρώσεις, δηλαδή τιμωρούνται οι γεωργοί για την κατάσταση αυτή όταν ούτως ή άλλως θα λήξουν οι ποσοστώσεις και γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια ζημία σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπήρξε υπέρβαση. Θα ήθελα η Τελική Προεδρία να παρουσιάσει μια σχετική πρόταση για το ζήτημα αυτό. Και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι έχουμε και το θέμα των χείρων που προέρχονται από την Αφρική Έχουμε τώρα αυτό το ζήτημα στην Πολωνία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη. Σε ένα-δύο χρόνια αυτό το πρόβλημα θα επεκταθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι θεμελιώδες να αντιμετωπίσουμε αυτή την όσο που διαδίδεται στην Ευρώπη από τους αφρικανικούς χείρους γιατί και η Λιθουανία έχει πρόβλημα και θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διατροφικής ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη θα ζητήσουμε από την Προεδρία να το αντιμετωπίσει. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριο Χόσλινγκ. Δύο λεπτά. Ευχαριστούμε για την επίσκεψη, κύριε Υπουργέ. Μπαίνω στα συγκεκριμένα θέματα. Αναφερθήκατε σε εμπορικές σχέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο νομίζω ότι κρίνονται από τους πολίτες εις ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Ε, δεν υπάρχει στις συμφωνίες που διαπραγματεύονται και εμείς οι βουλευτές ε, να εικάσουμε μόνο μπορούμε. Δεν μπορεί στο Διενικές να είναι σωστό αυτό τόσο σημαντικά θέματα να συζητούνται ε, με αποκλεισμό της κοινή γνώμης. Αυτό το επικρίνουν συνέχεια αλλά παρόλα αυτά δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να κάνουμε κάποιες σκέψεις επίσης ε, εν ώψη της κρίσης στο γεωργικό τομέα που δεν συνδέεται μόνο με το ρωσικό εμπάργο, αλλά στο γάλα ε, έχει προεκτάσεις. Δηλαδή πάλι η κρίση τώρα γίνεται συνειδητή σε όλους. Στο γάλα χρειαζόμαστε απαντήσεις. Τι θα γίνει μετά την ε, κατάργηση των ποσοστώσεων. Θα είναι σε ελεύθερη πτώση οι τιμές και αν δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις τότε θα ρίξουμε στην κρίση όλον αυτό το τομέα. Ε, Επίσης, ε, με το ρωσικό εμπάργο έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε εκείνους που αντιμετωπίζουν την κρίση, ιδιαίτερα τις γειτονικές χώρες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές αυτές. Πρέπει όμως να σκεφτούμε αν ο εξαγωγικός προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Γεωργίας ήταν ε, σωστός ε, γιατί είχαμε επενδύσει υπερβολικά πολύ στις εξαγωγές και δημιουργούνται εξαρτήσεις. Μιλήσατε για το... Ε, ε, ε και τους, ε, τις ανησυχίες των γεωργών σε αυτόν τον κλάδο. Θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα ούτω ώστε μέσα από τον νέο κανονισμό να καθησυχάσουμε τις ανησυχίες που υπάρχουν. Επίσης, παρά τις κρίσεις, πιστεύω ότι η προστασία του κλίματος δεν πρέπει να υποβαθμιστεί. Στην Γεωργία θα πρέπει το θέμα αυτό να συνεχίσει να έχει προτεραιότητα σε όλες τις σημασίες. Η Γεωργία και η προστασία του κλίματος είναι συνδεδεμένα εσένειες και τώρα και στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Σέντρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καταρχήν, να πω ότι το ρωσικό εμπάργκο έχει δείξει πως ε, έχει θεθεί σε κίνδυνο έχουν τεθεί σε κίνδυνο οι γεωργοί μα από τι πράξει Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και μόνο για να ευνοηθούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Επίση, βλέπουμε του κινδύνου μια κοινή γεωργική πολιτική, η οποία στι τελευταίε μεταρρυθμίσει ε, έχει προσανατολιστεί μόνο προ την εξαγωγή και εγκατέλειψε στην τύχη του ε, του ε, γεωργού που παράγουμε για την τοπική αγορά. Δεν είναι σοβαρή ούτε υπεύθυνη μια ΚΑΠ η οποία δεν θα σε προτεραιότητα την εσωτερική αγορά. Τώρα το παράδειγμα της απελευθέρωσης του συστήματος προσθέσεων στο γαλακτοκομικό τομέα νομίζω ότι επίσης ε, παρουσιάζει, παρουσιάζεται με αυτή την κρίση των τιμών που είχαμε ήδη πριν το ρωσικό εμπάργκο. Τρίτο, πιστεύουμε ότι οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών θα αποτελέσουν ένα ακόμα βήμα για την καταστροφή των Ευρωπαίων Γεωργών και της Γεωργίας. Δεν βλέπω στην παρουσίαση ε, του Ιταλού Υπουργού κανία πρόταση πραγματικής αλλαγής για μια πολιτική που να, λάβει, πράγματι υπόψη τα δικαιώματα και των καταναλωτών και των παραγωγών αλλά και, του περιβάλλον, εγώ θα ήθελα στην ε, εντολή σας να λάβετε υπόψη δύο θέματα. Να σταματήσετε τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών που ισχύουν επίση, ε, να μάθετε από τα διδάγματα, να υπάρξουν διδάγματα από όσα ζούμε και να υπάρξει μια νέα κοινή γεωργική πολιτική που να ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαίων γεωργών και όχι στα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών. Σας ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Καλό απόγευμα, κύριε Υπουργέ. Κάποια πράγματα να σας πω. Καταρχήν για τον έμπολα στη Δυτική Αφρική Τώρα όλοι το έχουν στο νου τους ή στις εφημερίδες τους ε, και ε, συνήθως ε, συνδέεται με φίδια ή επιθήκους κρέας που δεν τρώμε στην Ευρώπη, αλλά τρώνε οι Αφρικανοί. Εσείς θέλετε ότι έχετε συγκεκριμένο χορτοφυλάκιο εκεί και αν ε, ναι, στο Συμβούλιο των Υπουργών ε, θα ζητήσετε, θα πιέσετε για πιο συγκεκριμένες, πιο αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή, αν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει κάτι, τι θα γίνει παράλληλα και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, μπορείτε να πείτε ότι στην Ιταλία δεν θα κρατούνται πλέον οι οτόκες κότες σε κλοβούς και πρόκειται να ερευνήσετε τις φήμες που κυκλοφορούν ότι ε, χρησιμοποιούνται τέτοιοι κλοβοί και κλείνονται εκεί οτόκες κότες ε, σε πολύ μεγάλο νούμερα σε, στοιχείε σε κλοβών. Ευχαριστώ πολύ. Κατόπιν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό για να απαντήσει σε αυτές τις πρώτες παρατηρήσεις των συντονιστών. Και στη συνέχεια θα περάσουμε στις παρεμβάσεις των υπόλοιπων συναδέλφων. Για να πάμε τώρα στα κυρία σημεία, λέει ο κύριος Υπουργός, σε ό,τι αφορά το θεμελιώδες ζήτημα της ε, ε, εφαρμογής του νομοθετήματος δικαιώματα φύτευσης. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι η Προεδρία θα φροντίσει να γίνει σεβαστή η πολιτική συμφωνία που επετέχθη στο Κοινοβούλιο για το θέμα της διανομής γάλακτος και φρούτων στα σχολεία. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν. Δηλαδή ότι συζητούμε για μια πρωτοβουλία που θα έχει παιδαγωγική ε, αξία κυρίως ε, και θέλουμε να επικεντρωθούμε στην προσέγγιση αυτή για το θέμα των διαπραγματεύσεων ε, και κυρίως ε, για την TTIP, για την εταιρική σχέση, για την δικαιωτική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων, θα πρέπει να δούμε στην πραγματικότητα τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτή η συμφωνία για την Ευρώπη και φυσικά να μην ε, ξεχνάμε και τις επικρίσεις και τις προβληματικές πτυχές. Αλλά θα πρέπει να θέσουμε ψηλά τον πύχη για να ε, κάνουμε μία δουλειά, να παρουσιάσουμε προτάσεις για το θέμα αυτό και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για όλη την Ευρώπη από μια τέτοια στρατηγική σχέση. Ε, φυσικά υπάρχουν και προβληματικές πτυχές, ε, δεν τις ξεχνώ, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία είναι μια ευκαιρία και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα εξελίξουμε τα θετικά στοιχεία. Τώρα για το θέμα του χάλακτός. Όπως ε, ε, είπα, θα δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στο γαλακτοκομικό τομέα, κυρίως επειδή θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις από το 2015. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθούμε την αγορά και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει το ρωσικό εμπάργκο στις επιχειρήσεις μας, τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Το κάναμε αυτό όλο τον Αύγουστο σε συνεργασία με την Κομισιόν και πράγματι ε, ήρθαμε και σε μια πρώτη επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ήδη κατάλληλα εργαλεία που έχουν ενεργοποιηθεί. Θεωρώ ότι όλο αυτό το ποκέτο παρακολουθείτε και θα το διαχειριζόμαστε και τις επόμενες ημέρες. Για να δούμε, φυσικά θα έχουμε και κατά νου πώς μπορεί να βελτιωθεί. Κανείς δεν πιστεύει ότι όλα έχουν λήξει με τα νομοθετήματα και τις διατάξεις που έχουν εκπονηθεί μέχρι εδώ. Και εγώ θα ήθελα να εγγυηθώ ότι θα υπάρχει παρακολούθηση κατάσταση και αξιολόγηση βήμα το βήμα όλων ε, των εργαλείων που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν για να υποστηρίξουμε τι επιχειρήσει μα. Και αυτή είναι ε, φυσικά και η προσέγγιση που κρατήσαμε, που παρουσιάσαμε απέναντι στην Επιτροπή και τον Επίτροπο από την πρώτη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση που τέθηκε για το θέμα των σπόρων, θέλω να πω το εξής για το θέμα αυτό η Ιταλική Προεδρία λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται από το Κοινοβούλιο. Όμως ε, η Κομισιόν θα παρουσιάσει ένα νέο κείμενο και μόνο τότε έχουμε προβλέψει να προχωρήσουμε τις συζητήσεις της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου, λαμβάνοντας φυσικά και υπόψη τις ανησυχίε των ενστάσεων προέρχονται από το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Και νομίζω τα κάλυψα όλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Τώρα, δίνω το λόγο στους βουλευτές, ο κύριος Μπονάνο, ένα λεπτό κάθε ομιλητής τώρα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Εσείς αναφερθήκατε στους νέους γεωργούς, τους οποίους θα πρέπει να βοηθήσουμε. Εδώ είμαι, κύριε Πρόεδρε, είμαι μικρός όμως. Με καθυστερεί ο κύριος Ταραμπέλα, λέει Είχαμε ένα πολύ κακό παράδειγμα σήμερα το πρωί. Υπέβαλα μια προφορική τροπολογία υπέρ του ρυζιού και για γραφειοκρατικούς λόγους τελικώς βρεθήκαμε αντί για υπερασπιστές της Ευρώπης να ε, ε καθυστερούμε και να κολυσιοργούμε γιατί αντί να κάνουμε κάτι υπέρ στους... Ε, ε, για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Ε, κάναμε χάρη στους, ε, στους κατοίκους της Καμπότζης και στους Κινέζους που κάνουν ρίζια. Πραγματικά εγώ ήρθα εδώ και θέλω να κάνω κάτι για το ρύζι γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως Ευρωπαίους ενώ στην πραγματικότητα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Καμπότζης και της Κίνας. Είμαστε βλάκες εντός εισαγωγικών, ε, διότι εάν δαπανούμε τόσα εκατομμύρια ευρώ και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους γεωργούς οι οποίοι πλήττονται από το ρωσικό εμπάργο, πραγματικά πρόκειται για χρήματα τα οποία πετάμε και σκορπάμε, διότι αν είχαμε διαφορετική πολιτική με τη Ρωσία και τον Πούτιν θα είχαμε εξοικονομήσει χρήματα και θα υπήρχε και περισσότερη δουλειά για όλους. Εάν λοιπόν αυτή είναι η ιδέα της Ευρώπης, ε, ε, τι να σας πω. Διακόπτει ο πρόεδρο τον ομιλητή. Ο κύριος Κονίτ, κυρία Σκονίτ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά, γιατί δεν έχει διερμηνία στα λετωνικά. Οι Ευρωπαίοι γεωργοί επλήγησαν σκληρά από το ρωσικό εμπάργκο και Ιδιαίτερα στο γαλακτοκομικό τομέα υπάρχει πρόβλημα γιατί οι τιμές έπεσαν κατά 30-40%. Αν κάνουμε ε, την αναγωγή σε τιμή είναι 19 cents το λίτρο. Δηλαδή κάτω από το κόστος παραγωγής. Επίσης ε, οι εταιρείες γαλακτοπαραγωγής πλήττονται γιατί έκλεισε η ρωσική αγορά. Οι Λετονοί γεωργοί ε, χρησιμοποίησαν το 99,1% των ε, ποσοστώσεων. Και βέβαια δεν είναι μηχανή η αγελάδα, δεν μπορείς να τη σταματήσεις ε, να την αρμέγεις. Συνεχίζει να παράγει γάλα. Γι' αυτό ζητώ από το Ευρωπαϊκό το, το Συμβούλιο Γεωργίας να αποφασίσει να μην τιμωρήσει τους ε, γεωργούς που ξεπέρασαν τις ποσοστώσεις. Δεν είναι οικονομική μόνο η απόφαση, είναι και πολιτική απόφαση δεδομένης αυτής της καταστροφής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ναι, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Λίγα θα σας πω για το γάλα, συμφωνώ μαζί σας, αλλά νομίζω ότι είναι ε, προβλέψιμα τα όλα όσα θα συμβούν όταν σταματήσουν οι ποσοστώσεις οι πιο ευνοϊκές περιοχές θα είναι ωφελημένες και αυτές οι οποίες είναι πιο δύσκολες, οι ορεινές περιοχές και οι περιοχές της υπαίθρου θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Νομίζω το έχει συζητήσει αυτό και το Κοινοβούλιο και επομένως έχει προτείνει και ε, κάποιες λύσεις οι οποίες κατά την άποψή μου πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εγκριθούν διότι δεν αρκεί απλώς και μόνο η παρακολούθηση της κατάστασης. Θα ήθελα όμως να πιστήσω την προσοχή σας σε κάτι άλλο. Τους επόμενους μήνες και στην περίοδο της Ιταλικής Προεδρίας ε, θα υπάρξουν ε, σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο ICAN για την προστασία των ε, domain στο διαδίκτυο για πολύ σημαντικές ενδείξεις όπως για παράδειγμα το .wine, .n και διάφορα άλλα. Η Προεδρία ασχολείται με αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα διότι έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν ασχολείται, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα πράγματα τα αφήνουμε στη μοίρα τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπράνεν. Ευχαριστώ. αναφέρομαι σε αυτό που είπε στην αρχή ο Πρόεδρος και θέλω να αναφερθώ και στην Φεντερίκα Μογκερίνη η οποία ε, διαδέχθηκε τη Λέδη Άστον στις ε, κεφαλής της εξωτερικές υποθέσεις. Έχετε καλές ε, σχέσεις και συνεργασία. Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική βέβαια δεν πρέπει να υπαγορεύεται από τη γεωργική πολιτική. Καλό θα ήταν όμως η εξωτερική πολιτική να ενημερώνεται από τη γεωργική πολιτική. Πράγμα που θα μας ε, επιτρέψετε εσείς να εξασφαλίσουμε. Ελπίζω. Ευχαριστώ. Η κυρία, η Ντότζ, μιλήσαμε λίγο για τον ε, γαλακτοκομικό τομέα και είπατε εν παρόδο, κύριε Υπουργέ, ότι θα παρακολουθήσετε την κατάσταση. Θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία εξ ονόματος ε, των παραγωγών και μεταποιητών στην Ιρλανδία. Ε, οι τιμές μειώθηκαν και ε, τελευταία κατά 6%. Ε, θα υπάρξει μια μεγάλη αναταραχή στον τομέα αυτό. Κατά 7% αυξήθηκε η παραγωγή, η ζήτηση δεν ακολουθεί και το ρωσικό εμπάργο ιδιαίτερα στην εκλογική μου περιφέρεια, στη Βόρεια Ιρλανδία, πλήττουν το βούτυρο και το τυρί πάρα πολύ. Και οπωσδήποτε αυτό θα καταλήξει σε αποκορυφωμένο γάλα το οποίο θα επιδεινώσει το πρόβλημα της τιμής. Ε, Παράλληλα έχουμε περιορισμό των ποσοστώσεων. Μέχρι τώρα τις παρεμβάσεις τις χαιρετήσαμε, αλλά δεν αρκούν. Η ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι ευπρόσδεκτη, οι τιμές παρέμβασης είναι πολύ χαμηλές και δεν αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στην αγορά. Πρέπει λοιπόν να δούμε επιστροφές επί των εξαγωγών και πρέπει να σκεφτούμε το αδιανόητο και να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με την, τα αποτελέσματα της κατάργησης των ε, ποσοστώσεων και για να διευκολύνουν και να έχουμε μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν το σύστημα ε, ανάλογα με την περίπτωση και όχι ένα σύστημα για όλους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν, για τον τομέα τη ζάχαρης, η μεταρρύθμιση του 2006 επετρέπωσαν διαρθρώσει σε επίπεδο ε, ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας ε, και είχαμε πολλές ε, χώρες ε, λιγότερα αναπτυγμένες με τις χώρες ΑΚΕ, με χώρες των Βαλκανίων να συνάπτουν συμφωνίες για να εισαγάγεται εδώ, για να εισαγάγεται εδώ χιλιάδες τόνοι ζάχαρη και είχαμε πολλές αλλαγές. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο μαζικά πριν από τις ε, εκλογές αρνήθηκε το, η διάθεση στην ε, αγορά ε, του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, δηλαδή σπόρους, εμείς το απαρίψαμε αυτό. Ποια θα είναι η θέση της δικής σας Προεδρίας σε σχέση με το φάκελο αυτό. Θα συνεχίσει το Συμβούλιο αυτό το φάκελο ή θα απορριφθεί. Είναι σημαντικό για μας να ξέρουμε ποια θα είναι η θέση σας σε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, που τελειώσατε έγκαιρο. Ο κύριος Κουσμιουκ, κύριος μετά. Ευχαριστώ κύριε, Προ... Ε, κύριε Υπουργέ. Ε, δεν αναφερθήκατε στο ερώτημα του κυρίου Βοητσεχόφσκι, γιατί δηλαδή η Προεδρία μέχρι τώρα δεν επεχείρησε να κινητοποιήσει το αποθεματικό, το, το, το ταμείο που καλύπτει απώλειες στα πλαίσια της ΚΑΠ. Νομίζω ότι το εμπάργο πλήξε και τους 28 και τα 125 εκατομμύρια ευρώ που χρησιμοποιήσει η Κομισιόν όλοι ξέρουμε ότι δεν καλύπτουν επουδενή τις απώλειες ιδιαίτερα επειδή η αποζημίωση αφορά δύο περιπτώσεις ε, κυρίως. Δηλαδή, αν χρησιμοποιηθεί για φιλανθρωπικούς λόγους η καταστραφή εσοδεία. Και το πρόβλημα του εμπάργου είναι οι χαμηλές τιμές για όλα ουσιαστικά τα γεωργικά προϊόντα. Κάποια είναι ε, κάτω και από το κόστος παραγωγής τους. Ε, η χρησιμοποίηση μόνο αυτού του, η χρησιμοποίηση αυτού του αποθεματικού θα ήταν ε, καλή λύση για να αντιμετωπιστεί η, ε, το πρόβλημα. Ο επόμενος ομιλητής. Εσείς μάλιστα. Ευχαριστώ. Κατάγομαι από την Ιταλία, όπως και εσείς. Είμαι από τη Βενετία, μια περιοχή στην οποία ο αγροδιατροφικός τομέας είναι πολύ σημαντικός, αλλά από εσά ε, περιμένω κάποια συνέπεια την οποία δεν είδα εδώ, κάποια ακρίβεια. Φτάνει τα λόγια, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πράξεις. Τρία θέματα έχω να σας θέσω και ελπίζω να μας δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Καταρχάς, προάσπιση του αγροδιατροφικού τομέα όταν μιλάμε για τρόφιμα και λέμε πόσο καλά είναι τα προϊόντα μας και τα τραπέζια μας ε, ε, είναι αντικείμενο εισβολής από προϊόντα που έρχονται από όλες τις μεριές του κόσμου και δεν ξέρουμε πώς και πώς, ε, με ποιο τρόπο παράγονται και πού. Ε, τα, ταυτόχρονα η Ινδία μπλοκάρει τα κρασιά μας και τα γεωργικά μας προϊόντα λόγω ετικετοθεσίας προϊόντα εποχής, εποχικά προϊόντα τα οποία πλήττονται από άλλα ε, προβλήματα ε, χρειαζόμαστε πολύ ε, συγκεκριμένους ε, πόρους. Όσον αφορά το ρώσικο εμπάργο χρειαζόμαστε αποζημιώσεις διότι τα κονδύλια τα οποία δόθηκαν δεν αρκούν να αποζημιώσουν μόνο τη Βενετία και την περιοχή του Βένετο. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι άποψη έχετε εσείς, διότι ούτως ή άλλως έχει πληγεί ανεπανέρθωτα η γεωργία μας λόγω των παράλογων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Μόη, κύριε Υπουργέ, κάνετε μια ωραιότατη ομιλία αλλά ως συνήθω γεμάτο marketing, διαφημιστικά προϊόντα και καλά προϊόντα για την Ιταλική Προεδρία. Στην πραγματικότητα όμως η γεωργία στην Ιταλία είναι καταστροφική. Τι σκοπεύετε να κάνετε, κυρίω για να προστατεύσετε τη βιοπικιλότητα που είναι Ιταλική ε, και Ευρωπαϊκή κληρονομιά, ενώ εσείς είστε υπέρ της ε, απόλυτη έγκριση της TTIP. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να προστατέψετε τους γεωργούς και τους παραγωγούς της Νότιας Ευρώπης, οι οποίοι ε, δίνουν μάχη ενάντια στη συνθήκη που υπογράψατε εσείς για την εισαγωγή μαροκινών προϊόντων, τα οποία εισβάλλουν στις αγορέ μας με 0,15 σέντ το κιλό για τα προϊόντα μας και μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς κανέναν όλοχο για την ε, ποιότητα και την ποσότητα των φυτοφαρμάκων και μάλιστα οι γεωργοί ε, της Νότιας Ευρώπης Ευρώπης έχουν γονατίσει και δεν μπορούν ε, να ε, ξέρουν από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα και πώς μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν. Εσείς είστε υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση και τι σκοπεύετε να κάνετε για να τους προστατεύσετε. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω τι θέλετε να κάνετε για να προστατεύσετε από τις απάτες που έχουμε συνεχώς στην Ιταλία για τα εμβόλια, για την προστασία για διάφορες ε, ε ασθένειες φυτών και ζώων στην Ιταλία. Ευχαριστώ κύριο Σαμάτο και μετά ο Φλάνεγκαν. Η κυρία Νταμάτο. Καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για την ε, ε ελιά ε, και τα προβλήματα που υπάρχουν με το συγκεκριμένο βακτήριο το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών και επομένως θα πρέπει να γίνει εκρίζωση λόγω του γεγονότο ότι πλήττονται αυτέ οι ελιέ από το συγκεκριμένο βακτήριο. Αλλά εσεί κύριε Υπουργέ γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει ε, δυνατότητα. Διαπιστώθηκε ε, παρουσία κάποιων μικροοργανισμών, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη επιστημονική ένδειξη για την παρουσία του συγκεκριμένου βακτηρίου. Τι γίνεται λοιπόν με τα συγκεκριμένα μέτρα εκρίζωση. Πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη ει βάθο μελέτη, ανεξάρτητη μελέτη, που θα περιλαμβάνει και τη βοήθεια των γεωργών και την προστασία ε, συγκεκριμένων περιοχών. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση ε, που γίνεται ακόμα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά αν σκοπεύετε να ακολουθήσετε αυτή την άγουσα θα συνεχιστεί και άλλο. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξουν συγκεκριμένες ε, δραστηριότητες για να βοηθήσουν τα οικοσυστήματά μας, για να μπορέσουν να επανέλθουν στην ε, δύναμη που είχαν πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές και να ε, διαφυλάξουμε το μεσογειακό φυτό αυτό, την ελιά, και να προστατεύσουμε και το ελαιόλαδο από την απουλία. Ευχαριστώ. Ο κύριος και μετά ο κύριος Γιάρ σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά ξυλίας στην Ιρλανδία δόθηκαν στοιχεία ε, σχετικά με τη χειραγώγηση τιμών που αγνοήθηκαν, αναφέρθηκαν 125 εκατομμύρια ή 85 εν προκειμένου. Μπορείτε να λύσετε το θέμα ε, με τον Υπουργό μου όταν θα τον δείτε γιατί αυτό είναι πρόβλημα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν υπάρχουν ε, χειραγωγήσεις τιμών ή τέτοιες τέτοιοι πενιγμοί μπορεί να γίνει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν ε, ε, θέλουμε να, να, να ε, γίνουν τέτοιες επενδύσεις στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάρ και μετά κύριε Χάζελκαμπ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επαναλάβω τις ερωτήσεις, θα επαναλάβω μια πολύ σύντομη σε σχέση με την πτώση των τιμών λόγω του ρωσικού εμπάργου. Ε, το καλύτερο θα ήταν να αυξήσουμε την ενδοευρωπαϊκή κατανάλωση. Μιλήσαμε για τα προγράμματα στα σχολεία, γάλα και φρούτα. Δεν πιστεύετε ότι εν ώψη αυτής της κατάστασης ότι ήρθε η ώρα αυτά τα δύο προγράμματα να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα και να μειώσουμε την γραφειοκρατία, γιατί είναι πολύ γραφειοκρατικά και στη Γερμανία. Πολλά σχολεία γι' αυτό δεν χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε λίγο να σπάσουμε αυτές τις αλυσίδες, να αυξήσουμε την κατανάλωση και να απλουστεύσουμε το πρόγραμμα ώστε να καταναλώνονται περισσότερα ε, φρούτα και γάλα στα σχολεία. Ε, αυτό είναι μια πολύ σημαντική συμβολή στη μείωση της γραφειοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Χάζελκαμπ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Υπουργό για τη λεπτομερή παρουσίαση των προγραμμάτων. Δεν μιλήσατε όμως για την καλή μεταχείριση διαβίωση των ζώων, γιατί εκατομμύρια άνθρωποι προστατεύουν τα ζώα στην Ευρώπη και περιμένουν από εσά κάτι. Να αναφέρω κάτι. Κάθε μέρα βλέπουμε αυτά τα υπερφορτωμένα φορτηγά με ζώα από την Ολλανδία για παράδειγμα που ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη και έξω από την Ευρώπη και κάθε μέρα αυτά τα φορτηγά φορτώνονται με ζωντανούς χείρους που πάνε στην Ιταλία όπου θα γίνουν ε, μπέικον ε, και θα ξαναγυρίσουν στην Ολλανδία η, της Πάρμα στο προϊόν. Εμείς θέλουμε να φροντίσετε το θέμα αυτό της καλής διαβίωσης, χρόνη μεταφοράς, ζών των ζώων και άλλους κανονισμούς να λάβετε που θα προάγουν την καλή διαβίωσή τους. Ευχαριστώ ε, κύριε Ροπέ. Ο κύριος Ο κύριος Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ε, είναι κρίμα που δεν απαντήσατε το ερώτημα του Πολωνού συναδέλφου για τον Οθόδη. Είναι σημαντικό υποθέτω το ερώτημα. Ε, ε, την πανόλη των χείρων. Γιατί έκλεισε πρόσφατα ένα, μια μεγάλη εκμετάλλευση λόγω του, της πανόλης των χείρων και εσφάγησαν πολλά ζώα. Είναι πολύ ισχυρό το πλήγμα και ζωφερό το μέλλον. Η Ρωσία απαγόρευσε τις εισαγωγές ε, χειρίου κρέατος από τη Λιθουανία. Ακόμα και οι αγριόχειροι που ε, έχουν, έχουν ε, προσβληθεί και εισάγονται από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία και έχουμε καινούριε πηγές ε, μόλυνσης. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Γίνονται πολλές εικασίες σχετικά με την προέλευση της αφρικανικής πανόλης των χείρων. Ίσως έχει να ε, προέρχεται από τις ζωοτροφές, να μην οφείλεται μόνο στους αγριόχειρους. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό και να ληφθούν και μέτρα πρόληψης, γιατί το πρόβλημα αλλιώς θα αυξάνεται συνεχώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας ε, σε σχέση με την Ισπανική αίτηση να διευρυνθεί το καθεστώς ενίσχυσης για τη διανομή φρούτων και γαλακτός της ασφαλεία στο ε, λάδι και στις επιτραπέζιες ελιές. Δεύτερον, θεωρώ κατεπήγον η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να εφαρμόσει τη διεύρεση των ε, ενισχύσεων σε τομείς που θα ξεκινήσουν ε, την περίοδο διάθεσης και κυρίως αναφέρομαι στα εσπεριδοειδή που έχουν φυγεί ε, πάρα πολύ από το ρωσικό εμπάργκο θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί την το άνοιγμα νέων αγορών σε τρίτες χώρες ε, και την εξέλιψη των φυτογενομικών εμποδίων όπως αυτών που τίθενται από τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, για να ε, μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε την κατάσταση και επίσης θα έπρεπε να ληφθούν και νέες πρωτοβουλίες κατά της Ρωσίας ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού εμπορίου και να υπάρξουν και ευρωπαϊκές εκστρατείες προώθησης των πρόοδων που έχουν πληγεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε τρία σημεία, λέει η κυρία Γκυλερία. Είπατε αυτή θα αναθεωρήσετε ε, την Ευρωπαϊκή Στρατική 2020. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, η συμμετοχή των νέων στη Γεωργία. Νομίζω ότι δεν λύθηκε αυτό με τη μεταρρυθμιστικά. ΚΑΠ. Πρέπει να εμβαθύνουμε. Δεύτερη πτυχή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της ε, συμφωνίας σύνδεσης με τρίτες χώρες, γιατί ποτέ δεν ε, λαμβάνονται υπόψη ο αντίκτυπος ο πολύ συντριπτικός αντίκτυπος που υπάρχει σε όλη την ε, περιοχή. Εγώ προέρχομαι από την Ανδελουσία και συμφωνία με το Μαρόκο έχει πλήξει ιδιαίτερα την περιοχή μου. λοιπόν, ε, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να προτείνονται αντισταθμιστικά μέτρα, μέτρα αποζημίωσης για το θέμα της Ρωσίας. Ε, ποιο κανονισμό έχει προτείνει η Κομισιόν. Ο κανονισμός αυτός έχει αφήσει πολύ σημαντικά προϊόντα εκτός όπως το καρπούζι και το πεπόνι. Και αναφέρθηκε και ο κύριος Βελκάσερ, τα εσπερινδύει, τι θα γίνει με το κολοκυθάκι, με τη μελιτζάνα και να πω ότι υπάρχουν συνέπειες σε όλες τις οπορεκυπευτικές παραγωγές. Έτσι λοιπόν δεν φτάνουν τα χρήματα και ε, νομίζω ότι και η ημερομηνία της 30ης Νοεμβρίου είναι ένα μεγάλο λάθος. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω. Να σας δώσω το λόγο μάλλον, να πάρτε το λόγο. Θα είμαι ιδιαίτερα συνθετικός ε, για το ρύζι. Να πω ότι όλο το Συμβούλιο Υπουργών δίνει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό. Το συζητήσαμε το συγκεκριμένο θέμα τις ε, περασμένες ε, εβδομάδες, δική μας πρωτοβουλία και όχι μόνο. Ζητήσαμε από την Κομισιόν όχι μόνο να παρακολουθήσει με προσοχή την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά θέσαμε και το θέμα και προτείναμε η Κομισιόν να μελετήσει συγκεκριμένα την ενεργοποίηση της ρήτρα διασφάλισης. Ολοκληρώνουμε αυτό το φάκελο και για μένα είναι πρωταρχική σημασία σας, σημασία σας διαβεβαιώ. Τώρα, σας ευχαριστώ ε, που θέσατε αυτό το θέμα. Προσπαθήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ε, να συζητήσουμε και να θέσουμε στην ημερησία διάταξη με την Κομισιόν από τον περασμένο Ιούλιο το θέμα ε, της ε, ιδιοκτησίας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλά στο μέτωπο αυτό. Ελπίζω να υπάρχουν βήματα προς τον μπρος, γιατί νομίζω ότι είναι ένα μέτωπο για τα domain names. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρώπη. Τώρα για την Αφρική Πανόλη των Χείρων. Σας διαβεβαιώ ότι η Τελική Προεδρία θα προσδώσει ιδιαίτερη σημασία, μέγιστη σημασία. Θα συζητήσουμε και με τον Επιτροπό Μπόργκ τις επόμενες μέρες και όχι μόνο. Και υπόθεση αυτή την έχουμε παρακολουθήσει και τον Αύγουστο στις τελευταίες εβδομάδες όμως ε, να αναφερθώ και σε εσά που αναφερθήκατε στο θέμα του βακτηρίου της ξυλέλα μπορώ να σας πω ότι εμείς ε, εργαζόμαστε στην Ιταλία για να μπορέσουμε να λάβουμε δράση έτσι ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος ε, στο διαχείριση αυτής της προβληματικής για το θέμα του γάλακτος. Αναφέρθηκε πολλές φορές η λεπτή φύση του θέματος. Το πακέτο του γάλακτος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, θα ήθελα να υπενθυμίσω, σε διάφορα επίπεδα για τη βελτίωση της διαχείρισης και της λειτουργίας του κλάδου. Θα πρέπει συγκεκριμένα να καταφέρουμε να κάνουμε κάποια βήματα και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για να κατανοήσουμε πώς θα εξοπλιστούμε για να διαχειριστούμε αυτή την ευκαιρία. Ίσως ε, θα έπρεπε να δούμε τι συμβαίνει σε συγκεκριμένες περιοχές, αναφέρομαι στις ορεινές ε, και απομακρυσμένες περιοχές και στο δεύτερο και στον πρώτο πυλώνα ε, προβλέπονται κάποιε ενισχύσει, θα πρέπει να δούμε πώ η κάθε χώρα θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Και στην εθνική εφαρμογή αυτού του μέτρου εμείς ε, επικεντρωθήκαμε σε αυτό το θέμα. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας έδωσε η Νέα ΚΑΠ για το θέμα της ε, κρίσης με τη Ρωσία. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο που έχουμε κάνει μέχρι εδώ. Νομίζω ότι τις ε, προηγούμενες εβδομάδες εμείς ε, και με κάποιο γρήγορο τρόπο, με συνεννόηση με τους άλλους υπουργούς ε, και βάσει και της εμπειρίας της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας, προσπαθήσαμε να αρχίσουμε να τελειοποιούμε τα μέτρα. Και φυσικά Ζητήσαμε από την Κομισιόν και συγκεκριμένα μέτρα και για τα προκυπευτικά αλλά και για τα γαλακτοκομικά. Το πρώτο βήμα είναι αποθεματοποίηση για τα τυριά, το βούτυρο και τα γαλακτοκομικά. Εξελίσσεται τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή και σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και τις χρηματοοικονομικές διαθεσιμότητες. Εγώ μπορώ να πω ότι οι παρεμβάσεις Συνέφεραν ε, συνεισέφεραν ε, και στο θέμα των πόρων και των τρόπων και φυσικά την Παρασκευή με την Κομισιόν πρέπει να συζητήσουμε πώς βήμα το βήμα θα γίνει μια δουλειά που να ενισχύσει αυτά τα εργαλεία. Εγώ δεν θεωρώ ότι τόσο έχουμε κάνει μέχρι εδώ είναι κάτι που έχει ολοκληρωθεί, το είπαμε από την πρώτη στιγμή στην Κομισιόν, όμως θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από κάπου. Και εγώ νομίζω ότι ξεκινήσαμε με κάποια μέσα που μπορούν να μας βοηθήσουν. Φυσικά θα αναλύσουμε προσεκτικά την κατάσταση και θα πρέπει να διασταυρώσουμε κάποια στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να αναλάβουμε δράση και να αναπτύξουμε αποτελεσματικά εργαλεία εγώ δεν ε, θεωρώ ότι η παρακολούθηση είναι ε, κάτι στατικό ότι περιμένουμε για να ερμηνεύσουμε. Γιατί φυσικά θα πρέπει να προσφύσουμε τις επιχειρήσεις μας, όμως νομίζω ότι για να κάνουμε καλά τα πράγματα θα πρέπει να εξοπλιστούμε με τα κατάλληλα μέσα και ε, με τους συναδέλφους, υπουργού, την Περασκευή Θα είναι μια σημαντική συγκυρία το Συμβούλιο ε, φυσικά έχει ε, προωθήσει αυτό το ρεντεβού. Σας διαβεβαιώ ότι θα υπάρχει μια πολύ θετική σχέση με την κυρία Μικαρίνη. Ξέρω πόσο σοβαρή είναι και μπορώ να πω ότι αυτό που έγινε το Σάββατο δηλαδή όλο αυτό το θέμα που αφορούσε το ρωσικό εμπάρκο και το ευρωπαϊκό αγροτροφικό τομέα ε, μπορώ να πω ότι η κυρία Μικρίνη ήταν ενεργή και παρούσα και από το να Αύγουστο που είχε συγκληθεί το Συμβούλιο είχε οριστεί η συνεδρίαση της επόμενης Παρασκευής. Από την πρώτη στιγμή ως τελική προεδρία προσπαθήσαμε να έχουμε όλο αυτό το ενιαίο μέτωπο, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι συνέπειες στον αγροδιατροφικό τομέα. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στην εντέλεια με τη Φέντερ Καμικερίνη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμφωνία με το Μαρόκο που αναφέρθηκε, να υπενθυμίσω ότι ε, έχει συναυθεί εδώ και κάποιο καιρό. Ξέρουμε, γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες ε, του οποροκυπευτικού τομέα, όμως ε, πρόκειται για προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας ε, και είναι πιο πολιτικά. Δηλαδή, αν δούμε κάποιες προβληματικές, αν παρατηρήσουμε ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα, μπορούμε να έχουμε μια πιο, ένα πιο γενικό προβληματισμό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι μας ε, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί που πρέπει. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα. Μάλλον νομίζω ότι δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι απάντησα στα πιο σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. και η πληροφόρηση που σας δόθηκε και οι ερωτήσεις που ακούσατε θα σας βοηθήσουν για να, να θέσετε τα θέματα στο Συμβούλιο Υπουργών με τους ε, ομολόγους σας όσο καλύτερα τα στοιχεία, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, σας ευχόμεθα ό,τι καλύτερο και ευχαριστούμε και τους διερμηνείς, λέει ο πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, να, τους ευχαριστήσουμε δύο χειροκροτήματος. Και κύριε Υπουργέ, θα σας δούμε την επόμενη φορά μετά από την επιτυχή προεδρία που σας ευχόμεθα.